Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ε, πρωινή μας συνεδρίαση. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Ε, αφιερώσαμε πολύ χρόνο σε αυτή την επιτροπή και σε άλλες επιτροπές στην ε, προηγούμενη θητεία και εμπαθύναμε βεβαίως σε κάποια θέματα γιατί πρέπει να το παρακολουθήσαμε οπότε ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους ε, για το ότι μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε εις βάθος κάποιες πτυχές με την Κομισιόν. Και είναι κρίμα το ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν εκμεταλλεύονται την ευκαιρία να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες γιατί βεβαίως αυτό βοηθάει στο να λαμβάνετε μια σωστότερη απόφαση. Χαιρετίζω τους εκπροσώπους Κομισιόν, κυρίως τον κύριο Γούλμοντ ε, και τους δύο συναδέλφους και βεβαίως θα απαντήσετε στις γραπτές μας ερωτήσεις και θα έχουμε δυνατότητα μετά να επανέλθουμε. Κύριε Γούλμοντ, παρακαλώ έχετε τον, τον λόγο. Να, δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ που μας ε, δέχεστε εδώ πέρα, τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Βλέπετε πώς εκπροσωπούνται και οι δύο γενικές διευθύνσεις επιχειρήσεων και περιβάλλοντος, γιατί είναι κοινό μας έργο το να λειτουργήσει το ΡΙΤΣ. Κύριε Πρόεδρε, προφοριακά, καλό θα νομίζω να με αφήσετε να κάνω μια γενική παρουσίασαν σας στο πλαίσιο του που βρισκόμαστε. Ξέρετε πως ο Αντιπρόεδρος ο Ταγιάννη και ο Επίτροπος ο κ. πήγαν στο Ελσίνκι να τονίσουν την σημασία του ΡΙΤΣ και της υπηρεσίας βεβαίω, της υπηρεσίας της ΕΚΑ και να τονίσουν πως από 1η Δεκεμβρίου η ημερομηνία καταγραφής ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κατά το οποίο τόνισαν ε, σε πολιτικό επίπεδο και οι δύο τους ταυτόχρονα. Για τον λόγο αυτό έχουμε στη μία ομάδα των τριών θεσμικών οργάνων της Επιτροπής ε, της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας και της Βιομηχανίας ε, σε μια ομάδα επαφής διευθυντών όπως την λέμε για να δούμε ποια θα μπορούσαν να είναι τα προβλήματα για την καταγραφή, να καθίσουν όλοι μαζί και να βρουν λύσεις εντός ε, του νομικού πλαισίου του ΡΙΤΣ. Οπότε ήταν ένας ρεαλιστικός τρόπος ε, για να βρούμε λύσεις έτσι ώστε και η βιομηχανία και εμείς και η αποκεντρωμένη υπηρεσία να μπορέσουμε να σεβαστούμε την ε, προθεσμία της 1ης Δεκεμβρίου. Οφείλω να πω πως ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. 27 ζητήματα επισημάναμε ως πιθανώς προβληματικά όταν ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο έχουν όλα λυθεί, κάτι το οποίο βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα η δουλειά συνεχίζεται ομαλά. Είχαμε βεβαίω ε, στο τελευταίο κομμάτι ερωτήσεις από τους χρήστες, κάτι το οποίο αναφέρατε και στις ερωτήσεις σας οργανώσαμε από πλευράς Κομισιόν στο ίδιο πλαίσιο στην ομάδα των διευθυντών μία συνάντηση με αυτούς τους εκπροσώπους και την αποκεντρωμένη υπηρεσία, μια πολύ επικοδομητική συνάντηση και προσπαθήσαμε να βρούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι τα βασικά προβλήματα για αυτούς, γιατί όπως φαντάζεστε είναι δύσκολο να βρεθεί στο πλαίσιο αυτό να βρεθούν τα πραγματικά ερωτήματα, αλλά είμαστε όλοι ανοιχτοί ως, το, προς το να βρεθούν λύσεις. Θα δείτε λοιπόν τις λύσεις αυτές ε, στο site ε, της υπηρεσίας, οπότε μεταφράστηκαν αυτομάτως σε πολιτική. Η βιομηχανία Όσοι δεν ήταν δηλαδή συναντήσεις μας μπορούν να δουν εκεί πέρα πώς θα προχωρήσει η διαδικασία και σε τελική ανάλυση νομίζω πως ήταν μια καλή συνεργασία μεταξύ κομισιών της υπηρεσίας αυτής και της βιομηχανίας για να μπορέσουμε να είμαστε επιτυχείς την 1η Δεκεμβρίου. Αυτό το πλαίσιο ήθελα να, να θέσω στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ποιο θα συνεχίσει. Κάποιε από τι πρώτε ερωτήσεις θα τι δεχτώ εγώ και μετά θα αναλάβει ο κύριος Γουίλμοντ. Είχαμε το πρώτο ερώτημα, δεν θα το διαβάσω. Θα σας πω τι προετοιμάσαμε. Φαίνεται, με βάση όσα εξηγήσαμε, ότι ε, η διαδικασία είναι έτοιμη για τις 3 ε, Νοεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Χημική, ο Ευρωπαϊκός Χημικός Φορέας, η ΕΚΑ είναι έτοιμη και από τις 25 Οκτωβρίου υπάρχουν 8.500 ντοσχέ τα οποία είδαμε. Εμείς περιμένουμε 18.000 φακέλους να έχουν εγγραφεί μέσα στα πλαίσια της ε, προθεσμίας. Από ό,τι φαίνεται οι υποβολές γίνονται όλο ένα και περισσότερες όσο φτάνουμε στην προθεσμία και οι 38.000 φάκελοι και μάλλον οι 18.000 ε, φάκελοι θα φτάσουν στις 25.000. Δεύτερο ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, ένας από τους βασικούς ε, στόχους του REACH είναι μέσα στα πλαίσια της, ε, των αλλαγών στις προμήθειες να υπάρξουν αλλαγές και η βιομηχανία χρειάζεται χρόνο. Άρα, τη στιγμή που έχουμε καταγεγραμμένες ουσίες, ε, ακολουθούμε μια κάταντη διαδικασία και χρειάζονται 6 με 12 μήνες για την έγκριση. Η καταγραφή είναι το αρχικό στάδιο έτσι ώστε να μπορέσουν οι βιομηχανίες να ανταποκριθούν και να μας κοινοποιήσουν τις διαδικασίες, που, ε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίσουν. Σε αυτή τη ε, βάση προσαρμογής εμείς είχαμε θετικό feedback από τις βιομηχανίες και τις ουσίες. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Άρα η Επιτροπή οργανώνει ένα ειδικό workshop. Ε, απαντήστε τη δεύτερη ερώτηση και μετά θα έχουμε ερωτήσεις. Όπως σας είπα, είχαμε ένα δεύτερο workshop στις 27 Σεπτεμβρίου είχαμε 13 ε, βιομηχανίες που εκπροσωπούν τους ε, καταντιχρήστες. Ακούσαμε πολύ, ε, με πολύ προσοχή τις ανησυχίες. Ξέρουμε ότι ορισμένοι παρασκευαστές μας δώσαν ενθαρρυντικά στοιχεία, δηλαδή δεν είχαμε αρνητικό feedback από τις εθνικές οργανώσεις και είχαμε πολύ καλή επικοινωνία στην αλυσίδα προμηθειών. Άρα οι χρήστες ε, χημικών μπορούν να ανταποκριθούν στα πλαίσια της προμήθειας. Ε, επίσης θεωρούμε ότι αν υπάρξει κάποια ε, ε ρήξη στη διαδικασία θα μπορούσαμε να την επιλύσουμε bona fide. Λοιπόν, τώρα υπήρχε ένα διαδικαστικό ερώτημα Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διαβάζει γραπτές ε, αντίσεις, πράγμα το οποίο είναι χάσιμο χρόνο της Επιτροπής και δεν βοηθάει τους συναδέλφους. Αν υπάρχουν γραπτές απαντήσεις νομίζω ότι θα έπρεπε εκ των προτέρων να μας έχουν δοθεί για να τις έχουμε εξετάσει και να μπορέσουμε να διατυπώσουμε επιπρόσθετες ερωτήσεις διότι αυτό είναι καταφανής χρόνου. δεν μπορώ να το αλλάξω τώρα αλλά θέλω να σημειώσετε ότι είμαι, είμαι δυσαρεστημένος λοιπόν σημειώνουμε και εγώ δεν μπορώ να, το, να κάνω τίποτα ε, κάναμε γραπτές ερωτήσεις ζητήσαμε απαντήσεις και τώρα απαντούνται Αυτές ήταν οι πρώτες δύο ερωτήσεις. Τι θα γίνει. Θα δούμε καταρχήν τις απαντήσεις και μετά να συζητήσουμε. Νομίζω ότι θα είναι πιο έξυπνο, οπότε σας παρακαλώ πολύ να προχωρήσετε για να προβούμε μετά σε ερωτήσεις. Βεβαίως είναι ε, μία κατάσταση που εξελίσσεται ραγδαία και αν μιλάμε για αριθμούς αυτό που θα σας έλεγα εχθές δεν μπορεί να, ενδεχομένως να μην ισχύει σήμερα. Δεύτερον, η βιομηχανία θα έπρεπε να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ κατασκευαστών και χρηστών κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί μία διακοπή και διατάραξη της αλυσίδας προμηθείας που δημιουργείται με την καταγραφή του Ρίτσου. Επίσης, η, ε, αξιολόγηση επιπτώσεων του ΡΙΤΣ η οποία έγινε σε συνεργασία με την ε, βιομηχανία ήταν ε, ε, σε, ε, κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 2,9 εκατομμύρια διότι η αξία θα ήταν υψηλότερη από το κόστος της εγγραφής και θα αλλάζανε οι επιπτώσεις μέσω των αλλαγών των αξιών. Αλλά δεν έχουμε καμία ε, ε, κανένα αποτέλεσμα και ε, ενδεχομένως ορισμένες ε, ε, αρχές θα μπορούσαν να, θεωρητικά να αποσυρθούν από την αγορά αλλά ε, δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει στον τομέα αυτό ασάφεια και ορισμένες ουσίες να αποσυρθούν διότι ορισμένοι χρήστες να ήθελαν να αναλάβουν το κόστος και θα έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένες σύμβουλες σε συγκεκριμένους χρήστες. Ε, η ομάδα των χρηστών ε, επίσης ε, πρέπει να λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις και να παρακολουθεί την ετοιμότητα όλων των εταιριών σε σχέση με την προθεσμία του 2010 κατά τρόπον ώστε να υπάρξει συμμόρφωση της βιομηχανίας και να ε, επιληθούν τα προβλήματα όταν προκύπτουν. Το επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θυμίζει την ε, ε, εμπειρία της πρώτης καταγραφής όπου υπήρξαν πολλές δυσκολίες και ε, προς αυτόν τον στόχο πρόκειται να κάνουμε μία σειρά μελετών η οποία ε, θα στηριχθούν από την ΕΚΑ η οποία θα αναφερθεί ε, στα πρακτικά θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή. Θα πρέπει να εξετάσουμε τα βασικά θέματα και να ε, ε, σεβαστούμε τις μελλοντικές προθεσμίες καταγραφής κατά τρόπον ώστε του χρόνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, αναλύσει τα μαθήματα που απεκόμισε και να καθορίσει την επόμενη προθεσμία. Επίσης το, γραφείο, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Χημικών, η ΕΚΑ δηλαδή, έχει ζητήσει να ενημερωθούν οι ουσίες που δεν υπάρχουν στον κατάλογό της κατά τρόπον ώστε να ε, υπάρξει μία επαφή μεταξύ ε, της βιομηχανίας και των ενδιαφερομένων κατά τρόπον ώστε μέχρι τέλος Οκτωβρίου να, υπάρξουν, ε, να υπάρξει ένας κατάλογος όλων των ουσιών που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες σε όλη την αλυσίδα προμηθειών χωρίς όμως να έχουμε τις αντιδράσεις των κατασκευαστών. Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται ε, για την ομάδα των διευθυντών και όπως σας είπα ε, υπήρξε μία ε, ομάδα επαφών διευθυντών που καταρτίστηκε με πολύ θετικά αποτελέσματα που μπόρεσαν να καλύψουν τα πλαίσια του REACH. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα μαθήματα που απεκόμισε ε, θα ε, εξετάσει πώς μπορεί να διευρύνει τη συμμετοχή για την παρακολούθηση άλλων φάσεων εφαρμογής για να μπορέσει ή στο μέλλον να συζητήσει τους τομείς όπου χρειάζεται συνέχιση διότι υπήρξε στενή συνεργασία και συνέβαλε ε, στο να υπάρχει καταγραφή ε, γέρος. 8 ε, όσον αφορά την ε, ημερομηνία εγγραφή στις 30 Οκτωβρίου που εκπνέει ε, θα χρειαστεί περισσότερο προσωπικό και η ΕΚΑ σκοπεύει να βελτιώσει τους καταλόγους, να τους ενημερώνει εγκαίρως και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑ ενημερώνετε τακτικά για αυτές τις εξελίξεις. θα προχωρήσω με το επόμενο ερώτημα 9 για, τους, ε, για τα ε, ε, δασμολογικά θέματα και βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα της ευθύνης των κρατών μελών και ε, ε, η εφαρμογή μέσα στα πλαίσια του γραφείου προβλέπει ότι ε, θα υπάρξει μία εναρμόνιση και το φόρουμ έχει δημιουργήσει μία ειδική ομάδα συνεργασίας με τα τελωνία και διατυπώσει ορισμένες συστάσεις στα εθνικά τελωνία για το πώς μπορούν να συμμορφωθούν στις διατάξεις του ΡΙΤΣ και όσον αφορά την πιστοποίηση και παρακολούθηση της αγοράς προβλέπονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις τελωνιακές ορχές. Όσον αφορά τη δέκατη ερώτηση της μικρομεσαίας επιχειρήσεις, η, η διάζουσα κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή του REACH ε, όσον αφορά τα τέλη και ε, τους όγκους διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία ευξημένη ανταλλαγή εμπειριών και ε, μας έχει βοηθήσει η εμπειρία που είχαμε αποκομίσει στις πρώτες φάσεις και τις οποίες διαβιβάσαμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Επίτροπος Γιάννη έχει τονίσει το θέμα αυτό και ε, ε, ζήτησε από τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμπράξουν ιδίως γιατί λύγει η προθεσμία για την πρώτη καταγραφή. Άλλωστε προβλέπουμε να υπάρξει ικανοποιητική εξυπηρέτηση μετά την προθεσμία του 2010 και έχουν ήδη δηλώσει οι χρήστες ότι εκτιμούν τις ε, υπηρεσίες των Help Desk. Ε, το ΕΚΟ λοιπόν ε, η ΕΚΑ είναι έτοιμη να συμπράξει, να βοηθήσει, να ερμηνεύσει τα κατευθύνσεις έγγραφα κατά τρόπον ώστε ε, να υπάρχει μία ενημέρωση του οδηγού καταγραφής ε, και μετάφραση στις 22 γλώσσες ε, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμορφωθούν στις ανάγκες και επιταγές του ΡΙΤΣ. Ε, προβλέπεται όλα αυτά να γίνουν με δίκαιο τρόπο, αλλά η δίκαιη αντιμετώπιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πρόβλημα μέχρι στιγμής, διότι ε, δεν ε, υπάρχει διάφανη απέτηση από πλευράς τελών που πρέπει να πληρωθούν και γι' αυτό έχουμε κάνει ένα έγγραφο ερωταπαντήσεων για να επιλύουμε τις διαφορές και ε, να ε, προχωρήσουμε. Και τέλος, όσον αφορά τις μεταφράσεις. Η ΕΚΑ έχει μεταφράσει πολλά έγγραφα και το πρόγραμμα για το 2011 προβλέπει ότι οι μεταφράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν όπως θα συνεχίσει και η αναζήτηση πόρων από το δημόσιο προς το παρόν όλα τα έγγραφα υπάρχουν αγγλικά, μεταφράζονται όμως και το 2011 θα γίνει μία μελέτη σκοπιμότητος για να βελτιωθεί η επικοινωνία με το γραφείο και να μεταφραστούν σε διάφορες γλώσσες όλα τα έγγραφα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τις απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα, όπως είπε και ο Τζαέλς ε, Τσίτσεστερ, να μας δώσετε τις γραπτές απαντήσεις για να τις μοιράσουμε αμέσως στους συναδέλφους για να έχουμε και μία βάση. Αλλά έχουμε και μισή ώρα τώρα για να επανέλθουμε με άλλες ερωτήσεις. Πρώτος λοιπόν ο κύριος Λάγκεν. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, πληροφορίες. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο τελευταίο κομμάτι όσον αφορά τις επιπτώσεις στις μικρές και μισές επιχειρήσεις. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που σχόλησε το Κοινοβούλιο, μια βασική μας τοποθέτηση, ότι οι μεγάλες χημικές επιχειρήσεις οπωσδήποτε έχουν δυνατότητες και οικονομικά μέσα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσει αυτές, αλλά οι μικρομεσαίες συχνά θα μπορούσαν ίσως να σταματήσουν να παράγουν κάποια προϊόντα γιατί το κόστος είναι μεγαλύτερο από το κέρδος το οποίο θα βγάζουν από αυτά τα προϊόντα και είπατε πως η κατανομή του κόστους δημιουργεί προβλήματα και θα οδηγηθείτε σε μια δικαιότερη αντιμετώπιση. Τι γίνεται με τις ε, συμπράξεις, γιατί οι κονσόρτσια συχνά κάνουν μεγάλες επιχειρήσεις και υπάρχουν ε, παραδείγματα μικρότερων επιχειρήσεων που συνασπίστηκαν έτσι. Και βεβαίως ειδικά οι μεσαίες επιχειρήσεις ε, αυτό το οποίο μας λένε είναι πως είναι τόσα πολλά τα έγγραφα, τόσες πολλές ε, σελίδες, μιλάμε για εγχειρίδια 7.000 σελίδων που δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέρα από τα μεταφραστικά ζητήματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Μάλιστα. Ε, υποθέτω πως θα απαντήσετε αμέσως ε, κύριε Γουλμότ. Ναι, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ε, αμφιβολία ότι το REACH αποτελεί πρόκληση. Ως προς τη συμμόρφωση, η ΕΚΑ καταβάλει προσπάθειες με έγγραφα προσανατολισμού ή συστάσεων. Βεβαίως ο καθένας θα διαβάσει τα στοιχεία που τον ενδιαφέρει. Δεν χρειάζεται να διαβάσει και τις 500 σελίδες. Βεβαίως η ΜΜΕ συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο. Είναι δύσκολο για αυτές να ε, διαπραγματευτούν με τις ε, μεγάλες, ε, μεγαλύτερες βιομηχανίες, τα SIFs. Γι' αυτό είναι και ο ρόλος της ΕΚΑ πολύ σημαντικός για τους κανόνες ανταγωνισμού. Άρα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στα SIFs θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν. Νομίζω ότι δεν έχω τίποτα άλλο να πω ως προς τις ΜΜΕ. Ευχαριστώ πολύ. Τσίτσεστερ. Έχω ένα ακόμα ερώτημα για τις ε, συμπράξεις. Υπάρχουν τέτοιες συμπράξεις ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή όχι. We don't have information on the leaders δεν έχουμε τα, τα στοιχεία αυτά μέσα στα πλαίσια των ε, κοινοπραξιών. Από όσο γνωρίζουμε, πρόκειται για μεγαλύτερες επιχειρήσεις με μεγάλες ε, τεχνικές δυνατότητες. Δεν μπορώ να σας πω κατά πόσο υπάρχουν μήμοι έψιλων ε, επικεφαλής κοινοπραξιών. Τσίτσεστερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Νόμιζα ότι τα γερμανικά μου είχαν βελτιωθεί κατά πολύ σε αντίθεση με τον ε, συνάδελφό μου, μάλλον ε, σεβόμενο στο συνάδελφό μου, τον κύριο Λάγκ. Γνωρίζει η Επιτροπή γιατί έχουμε θίξει αυτά τα ζητήματα. Γνωρίζετε τις σοβαρές ανησυχίες των βιομηχανιών, του τομέα της βιομηχανίας, πραγματικά διότι υπάρχει μία εποδός σε όλες τις απαντήσεις σας, δηλαδή ε, σαν να υπάρχει μία συγκαταβατικότητα ή έλλειψη κατανόησης. Αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Δεν έχει νόημα να μας διαβάσετε γραπτές απαντήσεις που θα μπορούσατε να μας είχετε διανύμει πριν από την συνεδρίαση. Νομίζω ότι αυτό δεν μας τιμά Απαντώντας στο ερώτημα υπαριθμών 1, είπατε 8.500 φάκελοι έχουν ε, εγγραφεί στην ΕΚΑ και είπατε ότι η ΕΚΑ μπορεί να διεκπαιρεώσει 38.000 φακέλους μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Όμως οι βιομηχανίες την 1η Δεκεμβρίου δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία σωρία ουσιών που είναι πολύ σημαντικές στη διαδικασία αυτή παρασκευής και δεν υπάρχουν υποκατάστατα τι, τι εννοείται. Και αυτό το χάσμα μεταξύ 8.000 και 38.000 πώς θα πληρωθεί. Δηλαδή μιλάμε για 5 εβδομάδες για ένα διάστημα πέντε εβδομάδων. Στο, ε, στην απάντηση στο ερώτημα 2 και σας διέκοψα, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, μιλήσατε ότι οι κάταντι χρήστε θα έχουν 6 με 12 μήνες να συμμορφωθούν. Αυτό σημαίνει ότι μετά την προθεσμία έχουν μία περίοδο χάριτος για να ε, μπορέσουν να ενσωματώσουν όλες τις ουσίες ή αν δεν έχουν ε, καταγραφεί ή εγγραφεί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Απαντώντας στο ερώτημα 3 δηλαδή ποια βήματα θα πρέπει, σε ποια βήματα θα πρέπει, ποια βήματα θα πρέπει να προωθήσει η βιομηχανία έτσι ώστε να μην υπάρχει ρήξη στη διαδικασία. Είπατε ότι η διευθυντική ομάδα έδωσε εν μέρη μία απάντηση. Δεν μας δώσατε όμως απάντηση. Αυτό δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει. Εάν εγώ εκπροσωπούσα τη βιομηχανία, δηλαδή αν ήμουν βιομήχανος και έπρεπε να συμμορφωθώ σε πέντε εβδομάδες, αυτό δεν θα με έβρισκε σύμφωνο. Στο πέντε είπατε ότι υπάρχουν μελέτες εφαρμογής για του χρόνου, δηλαδή μετά την λήξη της προθεσμίας, όταν θα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και θα μπορούσα να συνεχίσω τέλος θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου ότι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από την έγκριση της νομοθετικής πράξης έχουμε αυτό το έγγραφο μόνο στα αγγλικά, μα μόνο στα αγγλικά. Μα αυτό τι να σας πω, είναι με εκπλήσει. Νομίζω ότι δεν μπορέσατε εσείς να συμμορφωθείτε αντιλαμβάνεστε τον, επί, τον κατεπήγοντα χαρακτήρα του θέματος. Γιατί ε, ε, μιλάμε για μεγάλες βιομηχανίες όπως την Airbus και στην ουσία εσείς αποτελείτε τροχοπέδι απαντώντας κατά αυτό τον τρόπο στις ε, ερωτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζετε την φύση του προβλήματος. Ναι, θα απαντήσετε θα απαντήσουμε μαζί. προς τον κύριο βουλευτή. Όχι, δεν υπάρχει κανένας ευσυχασμό. Αυτό το οποίο θα σα έλεγα είναι ότι για τον λόγο αυτό η ομάδα των ε, διευθυντών στην οποία συμμετέχει η Κομισιόν, η Αποκεντρωμένη Υπηρεσία και η Βιομηχανία ξεκίνησαν δουλεύει πριν από πολλούς μήνες. Η ομάδα αυτή επεσήμανε τα προβλήματα και συνεργαζόμαστε με τη βιομηχανία για να βρούμε λύσεις, τις λύσεις που ζητούσε η βιομηχανία. Οι λύσεις δημοσιεύονται. Οπότε για αυτό το οποίο ρωτήσατε πώς θα ξέρουν οι άλλοι ποιες λύσεις ε, βρίσκονται, δημοσιεύονται αυτά από την ε, υπηρεσία. Τι λύσεις βρίσκουμε και ρεαλιστικά με ποιον τρόπο μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας ευησυχασμός, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά τους τελευταίους 7 μήνες. Είμαστε σε επαφή με τη βιομηχανία και μέχρι στιγμής η βιομηχανία μας λέει πως όλοι κάνουν ό,τι μπορούν και από εκεί, σε αυτά βασιζόμαστε. Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερε πληροφορίε από αυτέ που μας δίνουν για τους χρήστε προς τα κατάντη. Αυτομάτως μόλι προέκυψαν ε, ερωτήματα ήρθαμε σε επαφή με αυτό το κλάδο τη βιομηχανία. Προσπαθούμε και μαζί τους αποτελεσματικά να λύσουμε το πρόβλημα ή να απαντήσουμε δηλαδή στις ερωτήσεις. Αλλά το πρόβλημα είναι εκεί πως είναι πολύ δύσκολο να δούμε πού βρίσκεται ακριβώ το πρόβλημα. Εάν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο στοιχείο στην αλυσίδα, πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε πού βρίσκεται. Είναι πιθανό πω θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά μπορεί να μην υπάρξει κιόλα. Οπότε συνεργαζόμαστε με τους χρήστες για να το δούμε αυτό και τις επόμενες μέρες και θα τους συμπεριλάβουμε και στην ομάδα αυτή των διευθυντών ε, κάτι το οποίο δεν γινόταν στο παρελθόν για να κάνουμε μια γενική συζήτηση μαζί τους. Αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση. Και ο Γκρέαμ νομίζω θέλει να συμπληρώσει κάτι. Ναι, να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα για τις ανησυχίες για τους ε, χρήστες ε, προς τα καταντή, όπως είπε και ο συνάδελφος, υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα για το ποιες ουσίες θα αποσυρθούν, εάν αποσυρθούν κάποιες και τι αποτελέσματα θα έχει αυτό. Βεβαίως αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τις επιχειρήσεις και μία ουσία να αποσυρθεί μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε αριθμό επιχειρήσεων. Δεν ξέρουμε πού χρησιμοποιούνται ακριβώς αυτές οι ουσίες και ποια οικονομική λειτουργία παίζουν. Οπότε γι' αυτό ακριβώς συνεργαζόμαστε στενά με τους χρήστες για να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Ιδεώδης λύση θα ήταν μια λύση η οποία δεν θα διέκοπτε καθόλου την παροχή του προϊόντος. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να υπερβούμε τον κανονισμό. Είμαστε εντός του νομικού πλαισίου. Εάν δεν γίνει αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ε, εργαζόμαστε εντατικά αλλά δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ποια θα είναι η λύση ούτε σε εσάς ούτε στους χρήστες. Για το... την μετάφραση του Reach IT. Ίσως η προηγούμενη μου απάντηση δεν ήταν αρκετά σαφής η τεκμηρίωση και οι σελίδες ε, στο διαδίκτυο, οι σελίδες βοήθειας έχουν μεταφραστεί, αλλά οι οθόνες του χρήστη όταν μπαίνει στο σύστημα δεν έχουν μεταφραστεί. Ε, όπως σας είπα η Κομισιόν ε, ζήτησε από την έκανα το μεταφράσει και η αποκεντρωμένη υπηρεσία θα κάνει μια αξιολόγηση του αν μπορεί να το κάνει. Επίση για του φακέλου. Οπωσδήποτε δεν υπάρχει ευσυχασμό, αλλά δεν ανησυχούμε και υπερβολικά γιατί η εμπειρία μας με τις προηγούμενες προθεσμίε ε, όσον αφορά την νομοθεσία χημικών ουσιών δείχνει πως ε, προς το τέλος υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση της εργασίας. Τέλος, για το ότι δεν ε, μοιράσαμε τις απαντήσεις μας. Ε, τις απαντήσεις μας τις αλλάζαμε ακόμα και τη στιγμή που καθόμασταν εδώ πέρα και ο πρόεδρος ξεκινούσε την συνεδρίαση. Οπωσδήποτε βεβαίω μετά τη συνεδρίαση θα σας δώσουμε τις απαντήσεις γραπτός. Ευχαριστώ. Επειδή ο χρόνος πιέζει τώρα θα ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις μαζί. Τζάιλς, αν θέλεις να επανέλθει και μετά θα δώσω λόγο και στους άλλους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ ο χρόνος είναι το ουσιώδες. Επτά μήνες πριν μας είπατε ότι συστάθηκε αυτή η ομάδα εργασίας. Αρκετά αργά δηλαδή εσείς ή η βιομηχανία συνειδητοποίησατε ότι υφίσταται πρόβλημα. Αυτό μου το ανέφεραν έξι εβδομάδες πριν, δηλαδή πολύ κοντά στην προθεσμία. Απελπιστικά κοντά. Εφόσον η νομοθεσία αυτή συστάθηκε πέντε χρόνια πριν, μπορείτε να μας πείτε γιατί αναλάβατε δράση τόσο αργά. Καταλαβαίνω ποιος είναι ο, ο βασικός στόχος και βεβαίως θέλετε να μάθετε να ρίξετε φως στις άγνωστες ουσίες, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε τόσο μικρή, μικρό χρονικό διάστημα. Κυρία Χέρτσοκ. Ευχαριστώ. Ε, επειδή ήμουν σκιώδης για το θέμα αυτό, μπορώ να σας πω ότι θα θέλαμε να επιτύχει το εγχείρημα, το εγχείρημα αλλά δεν είναι γραφειοκρατικής υφής. Εάν είναι γραπτές οι απαντήσεις και αν μιλάτε ε, για 40.000 ουσίες, τότε μπορείτε να απαντήσετε στις 7 ή 10 ερωτήσεις. Το REACH ε, δεν είναι γραφειοκρατικό εγχείρημα. Θέλαμε να δούμε ποιοι είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι. Βρήκατε που υπάρχουν αυτοί οι μεγάλοι κίνδυνοι και πού βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα. Γιατί εμείς είπαμε στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες ότι αυτό το αντίτιμο πρέπει να καταβάλλεται διότι υπάρχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Το άλλο ερώτημα έχει ως εξή. Μερικοί τα κατάφεραν, αλλά πόσα, ποιο ε, είναι το διακύβευμα και πόσοι χάθηκαν στο δρόμο. Διότι αυτό είναι ε, μεγάλο θέμα για χώρες που δεν έχουν μητρική γλώσσα στα τα αγγλικά. Εάν οι βιομηχανίες ε, πρέπει να μεταφράσουν αυτό το ε, κείμενο, τότε αυτό είναι άδικο για αυτές τις χώρες, τη στιγμή που δεν χρησιμοποιούν τα αγγλικά ως βασική γλώσσα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια γραπτή έκθεση σε όλες τις γλώσσες. Η ΕΚΑ ο κανονισμός αρκεί ή χρειάζεστε επιπρόσθετα στοιχεία που, στα οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί το Κοινοβούλιο ή νομίζετε ότι μπορείτε να το κάνετε. Τέλος, τι γνώμη έχετε για τους άλλους κανονισμούς. Ε, σε σχέση δηλαδή με τα βιοκτώνα και ούτω καθεξής. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε αποδυναμώνεται το ΡΙΤΣ Άρα μιλάμε για άλλες ουσίες τη στιγμή που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε το REACH. Αυτό αποδυναμώνει το έργο σας ή το ενισχύει. Νομίζω ότι αυτό αφορά όλες τις βιομηχανίες. Μιλάμε για μια βιομηχανική πολιτική. Αυτό είναι το επίκεντρο της πολιτικής. Ευχαριστώ. Ε, εγώ ήμουν ε, έτοιμος να ξεκινήσουμε σε 9 και 9 και 10 ήμασταν δύο, υπήρχαν μόνο δύο. Διότι στις 10 θα έχουμε άλλους συναδέλφους οι οποίοι θα έρθουν να ψηφίσουν και θέλουν η ψηφοφορία να γίνει εγκαίρως. Δεν μπορούν όλα να γίνονται σωστά εάν δεν καλύπτουμε τις προϋποθέσεις. Ο κύριος Ματσάουερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία του συστήματος καταγραφής αλλά και εγώ έχω ορισμένες ανησυχίες ε, παρόμοιες με αυτές που εξέφρασε ο κύριος Σίτσεστερ σχετικά με ε, το χρονοδιάγραμμα και ο κύριος Λάγγεν μίλησε για το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολική η επιβάρυνση των μικρομεσαίων ε, για τα διοικητικά θέματα. Ορισμένα δηλαδή προβλήματα ναι μεν έχουν επιληθεί αλλά ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται και ορισμένες ε, ουσίες θα μπορούσαν να αποσυρθούν στο μέλλον και άρα θα πρέπει να προβλέψουμε επαρκή χρόνο για αυτή τη διεργασία. Έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί σχετικά με την ε, περαιτέρω χρήση ζώων για τις ε, έρευνες. Πιστεύετε ότι η διαδικασία αυτή θα αυξήσει την χρήση των ζώων μπορεί να αντισταθμιστεί χρησιμοποιώντας ε, τα ισχύοντα στοιχεία με κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή ε, είχε να η εισηγήτρια για αυτό το θέμα, ανησύχησα τόσο πολύ, ώστε ε, πριν μία εβδομάδα είχα μία συνάντηση με έναν υπάλληλο του γραφείου. Οι δε απαντήσεις σας, ε, κατά τη γνώμη μου, είναι εν μέρη χρήσιμες και εν μέρη όχι. Και συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες. Δηλαδή, αυτή η νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντική για το περιβάλλον, για τους Ευρωπαίους και ιδίως για τις χώρες οι οποίες όντως δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα αυτό εις βάθος στο παρελθόν. Δεν θέλω ε, να αναφέρω κάποιο συγκεκριμένο ε, αλλά ο χρόνος από όταν ε, λήφθη η απόφαση μέχρι τώρα έπρεπε να επαρκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε πει ότι το χρονοδιάγραμμα ήταν ε, σωστό, ότι υπήρχε η οργάνωση με το σωστό τρόπο, είχε καταρτιστεί και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν προβλήματα που προκύπτουν και μπλοκάρουν το σύστημα. Η ερώτηση μου λοιπόν κύριε Πρόεδρε είναι καταρχήν ε, στην Άνοιξη θα ήθελα να ε, είμαι επικεφαλής μίας ε, αντιπροσωπείας να συζητήσω τα θέματα αυτά στο Ελσίνκι. Ελπίζω ότι θα το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών κατά τρόπον ώστε να δούμε πού προκύπτουν τα προβλήματα και πού υπάρχουν συμφορήσεις. Και το δεύτερο είναι τι κάνετε σχετικά με τις εμπλεκόμενες ε, επιχειρήσεις και τους υπευθύνους για να τους ενημερώσετε για το τι κάνετε. Ε, τους δίνετε και άλλες πληροφορίες ή πόσο προχωράτε. Διότι το να καταρτήσετε μία ομάδα και να έχει ένα όνομα δεν ε, σώνει την ε, συγκεκριμένη επιχείρηση, δηλαδή όσον αφορά τις μεμονωμένες επιχειρήσεις πώς τους ενημερώνετε, πώς μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους ασφαλώς. Κύριε Λισκόκ. Eh, Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εδώ το REACH ε, αντιπροσωπεύει την πιο ε, σημαντική ε, πρόοδο για τις χημικές ουσίες ασχέτως των συμφερόντων που είχαν εμπλακεί όταν υιοθετήσαμε αυτήν την νομοθεσία. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς πολλά συμφέροντα και εδώ εκπροσωπούνται πολύ δυναμικά αλλά η νομοθεσία είναι αρκετά καλή. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες ε, ασάφειες όσον αφορά τις ε, προθεσμίες ε, εγγραφής και αναρωτιόμαστε πώς οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να σεβαστούν αυτή την νομοθεσία. Η εντύπωσή μου και η εντύπωση της ομάδος μου είναι ότι ε, η ε, το γραφείο και οι επιχειρήσεις συνεργάζονται για να μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει και για τις μεγάλες και για τις μικρές επιχειρήσεις. Και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά εις ε, τις ανάγκες, η ομάδα επαφών και η ομάδα ε, συνεργασίας ε, τελικά αποβλέπει ε, στο να διευκολύνει την εργασία του Ρίτς. Βέβαια θα πρέπει η νομοθεσία να έχει εφαρμοστεί σωστά. Και θα ήθελα σαν ε, νομοθέτες να αναλάβουμε τις ε, ευθύνες μας και ε, να την στηρίξουμε κατά τρόπον ώστε όλα να λειτουργήσουν σωστά πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα. Πολλές φορές όμως διονγκώνουμε το πρόβλημα και έχουμε την εντύπωση τελικά ότι ορισμένοι θέλουν να υποθάλψουν αυτή την νομοθεσία για να μην εφαρμοστεί, το οποίο θα ήταν μια πολύ κακή ιδέα. Χρειαζόμαστε το ρίτς και ιδίω χρειαζόμαστε να είμαστε σύμφωνοι επί του γεγονότος ότι το ρίτς πρέπει να προχωρήσει και είναι καλή νομοθεσία. Ο κύριος Λάνιεν. Πρώτα απ' όλα, μας είπατε στις ε, απαντήσεις πως έχετε μεταφράσει τα έγγραφα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετά απαντήσατε στον κύριο Τσίτσιστερ πως έχετε μεταφράσει μέρος των εγγράφων, λίγο πριν λήξει η προθεσμία. Τι γίνεται εδώ πέρα, μας λέτε διαφορετικά πράγματα. Παλέψαμε χρόνια εδώ πέρα για να υπάρχει μια ίση μεταχείριση. Και τίθεται το ερώτημα, είναι η Κομισιόν διατεθειμένη και έτοιμη να προβεί σε παράταση της ε, προθεσμίας εάν δεν, υπάρχει, δηλαδή, εάν δεν υπάρχουν δίκαιες προϋποθέσεις για να έχουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση στις πληροφορίες. Μετά μας είπατε πως έχουμε σχέδια ανάγκης ε, και να αυξήσουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας μας κατά 400% στο τέλος ε, της προθεσμίας. 400%! Απορώ δηλαδή για το ότι δεν πρότεινε κανείς από εσά μια παράταση της προθεσμίας. Αυτή παρέμβαση. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Χέρτσοκ ότι θα πρέπει να διακρίνουμε το γλωσσικό. Τα αγγλικά είναι η γλώσσα του Σέξπιρ ε, και είναι διαφορετική η χρήση ως προς την ανάγνωση έργων του Σέξπιρ ή θεμάτων όπως το παρόν. Θα ήθελα να πω ότι είμαι απόλυτα απογοητευμένος γιατί είχαμε το σύστημα δοκιμών των χημικών ουσιών στο παρελθόν. Στη χώρα μου είχαμε έναν εθνικό οργανισμό δοκιμών για όλα τα προϊόντα, όλες τις ουσίες και σύμφωνα με τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταργήσαμε αυτό τον οργανισμό που λειτουργούσε πολύ καλά, οργανισμό δοκιμών ουσιών και προϊόντων. Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα δηλαδή ως προς τις ανάγκες των ε, καταναλωτών μας, των πελατών μας και των χρηστών, ως προς την προμήθεια της αγοράς. Ελπίζω να πληρωθεί αυτό το χάσμα στο μέλλον, αλλά είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί το σύστημα όπως είχε προταθεί από την ε, Κομισιόν δεν θα είναι απόλυτα λειτουργικό όπως θα έπρεπε. Ζητώ την κατανόηση. να, ε, ε, ε, να έχετε κατανόηση για να μπορέσουν να απαντήσουν για δύο λεπτά. Αγγέλικα Νίμπλερ, <coughs> δεν θα χρειαστώ καν δύο λεφτά. Ήθελα να στηρίξω τη σχόλια του κυρίου Λάγκεν διότι ήμουν εχθές ε, στη Βαβαρία ε, σε ένα χώρο που υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χημικές όπου αντιμετωπίζεται ένα τεράστιο πρόβλημα με όλα τα έγγραφα διότι υπάρχουν τα έγγραφα μόνο αγγλικά και αν δεν παραταθούν οι προθεσμίες και παρόλη την καλή θέληση όλων να καλύψουν τις προϋποθέσεις είναι αδύνατον. Δεν είναι δυνατόν να απαιτήσει κανείς από αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι όλοι οι επίτροποι μας λέγουν πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσει κανείς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό θα ήθελα και το ΡΙΤΣ να το αναγνωρίσει και να παρατείνει τις προθεσμίες. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή έχει πάλι το λόγο και αν συμφωνείτε πρότεινα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβλέποντας ότι πρέπει να ψηφίσουμε στις 10 και έρχονται ήδη όλοι οι συνάδελφοι να απαντήσει η Επιτροπή ήδη σε 5-6 ερωτήσεις. Δεν θα υπάρξουν όλες οι λεπτομερείς ε, απαντήσεις αλλά θα τις λάβουμε γραπτός και μετά θα χρειαστεί ενδεχομένως να επανέλθουμε διότι ενδεχομένως θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα πολλά θέματα. Πρώτη δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Ο κύριος Μπερμότ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, όλοι λέτε ότι το θέμα είναι σημαντικό. Τώρα θα ήθελα να προσέξετε τις απαντήσεις της Επιτροπής. Ευχαριστώ εντάχει. Το ερώτημα ήταν για τους κινδύνους. Έχουμε ανιχνεύσει κινδύνους. Ναι, έχουμε ανιχνεύσει κινδύνους διότι έχουμε αναγνωρίσει νέους κινδύνους κατά την εγγραφή. Γι' αυτό τα Μητρώα ανταποκρίνονται στόχους βελτίωσης της ασφάλειας. Βεβαίως μας απασχολούν οι ΜΜΕ. Έχετε δίκιο για τη μετάφραση. Θέλαμε η ΕΚΑ να συνεχίσει την εργασία της με τις ε, μεταφράσεις ε, έτσι ώστε να μεταφραστούν τα σημαντικά αυτά έγγραφα για τις ΜΜΕ μέσα στην προθεσμία. Τώρα, ως προς μεμονωμένες ε, ΜΜΕ δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή από τις Βρυξέλλες. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεων. Απλώς έχουμε, προωθούμε ε, συγκεκριμένες εκστρατείες μέσα στα πλαίσια εκδηλώσεων αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε στις μεμονωμένες ΜΜΕ ως προς τις δοκιμές στα ζώα. Προσπαθούμε να μειώσουμε τις δοκιμές αυτές, αλλά ορισμένες επιπρόσθετες δοκιμές χρειάζονται οπωσδήποτε. Προσπαθούμε όμως να συρρυκνώσουμε αυτό το πλαίσιο, να μειώσουμε δηλαδή αυτές τις δοκιμές. Η ΕΚΑ χρειάζεται ε, περισσότερη υποστήριξη. Μπορέσαμε να βρούμε ε, περισσότερους πόρους εάν χρειαστούν για τις εγγραφές κατά 400%. Γιατί συστάθηκε η DCG φέτος. Η ομάδα, η ομάδα των διευθυντών φέτος. Γιατί χρειάστηκε να δούμε ορισμένα ζητήματα επιγόντως. Ε, ως ε, προς τις παράπλευρες απώλειες ή τις κύριες απώλειες. Δεν βρήκαμε πτώματα στους δρόμους ακόμα, αλλά θα γίνουν μελέτες του χρόνου για να δούμε τις επιπτώσεις στην αγορά. Και ελπίζουμε να μην ε, έχουμε μεγάλες απώλειες του χρόνου, αλλά θα το δούμε μεταξύ των άλλων επιπτώσεων του Ριτς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Τα άλλα ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν μέχρι στιγμής θα απαντηθούν γραπτός. Ε, λέγω λοιπόν καταρχήν στην ε, Επιτροπή ότι την ευχαριστώ, θα επανέλθει, θα χρειαστεί να επανακάμψει διότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα του γεγονότος ότι εχθές ε, όπως συζητήσαμε εχθές οι ε, επιπτώσεις ε, των νομοθεσιών καταρχήν δεν είναι πάντοτε σαφείς πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι έχουμε αποφασίσει και τι προβλήματα προκύπτουν στη συνέχεια, τι περιπλοκές Άρα θα πρέπει να είστε πιο ευέλικτοι από πλευράς χρόνου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προχωρήσετε με ένα θέμα το οποίο δεν καλύπτει το χρονοδιάγραμμα που χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα. Δηλαδή στην ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες σας μαζί για να ψηφίσουμε. Έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες σήμερα, οπότε σας παρακαλώ να δείξετε λίγη προσοχή και να με βοηθήσετε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θέλω λίγο τη βοήθειά σας και την προσοχή σας γιατί στην αρχή είναι απλά τα πράγματα, μετά υπάρχουν κάποιες πολύπλοκες ε, ψηφοφορίες. Κυρίε και κύριοι, η γραμματεία προσπάθησε να κάνει την ε, σειρά των ψηφοφοριών έτσι ώστε να τηρήσουμε όλους του Είναι λίγο περίπλοκο, αλλά αυτό θα κάνουμε δεύτερο, το οποίο θα ήθελα να διατυπώσω. Καμιά φορά Μπαίνω και εγώ στη θέση των απλών βουλευτών που δεν είναι συντονιστές ή εισηγητές. Είναι δύσκολο να σχηματίσει κανείς άποψη όταν λαμβάνει το προηγούμενο βράδυ ή το πρωί τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Απευθύνομαι σε όλους. Πρέπει να σκεφτούμε πώ θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα για να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Είναι σχεδόν αδύνατον να εξετάσει κανεί τα πράγματα. Κάποιοι, λίγοι, που είναι σκιώδεις ηγητές, συντονιστές κτλ. βεβαίως έχουν πιο ακριβή εικόνα. Αλλά συχνά οι υπόλοιποι συνάδελφοι δυσκολεύονται όπως και εγώ σήμερα. Περνάμε τώρα λοιπόν στην ψηφοφορία. Το πρώτο σημείο είναι το σημείο 9 που είναι απλό. Μιλάμε για σχέδιο έκθεση απλοποιημένη διαδικασία χωρίς συμφωνία Μιλάμε για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της κοινότητας και της Ιορδανίας. Ποιος συμφωνεί με αυτό. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο 10 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ιαπωνίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της Ουκρανίας υπέρ. Στοπ, σταματήστε κυρία Εκ. Συμφωνώ με το πόσο γρήγορα πάτε κύριε Πρόεδρε, αλλά πάρτε και καμία ανάσα μεταξύ των διαφόρων φακέλων για να μπορούμε να γυρίσουμε τις σελίδες. Okay. Yeah, yeah, yeah. Ε, εντάξει, ευχαριστώ. Τόσο, τόσο γρήγορα πήγαινα, συγγνώμη. Λοιπόν, τι θέλετε, πιο γρήγορα ή πιο αργά και τα δύο που μου λέτε δεν γίνονται. Λοιπόν, εντάξει, πιο αργά από ό,τι πριν. Ναι. Ωραία, Ουκρανία, ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Ευρωπαϊκή κοινότητα και νήσι Ποιο Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στα πιο δύσκολα. Σημείο 13, ενεργειακή στρατηγική. Μια στιγμούλα παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα να βρω και εγώ τη σελίδα. Ποιος θέλει πρώτος τον λόγο. Η κυρία Εκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως συντονίστρια συζήτησα και εγώ με του άλλου στον κατάλογο των ψηφοφοριών να την προσοχή σας στις ε, συμβαστικές προτάσεις 27α και β. Εγώ, κύριος Ρόντε και Χατζημαρκάκης έχουμε την τροπολογία 239 που ζητήσαμε να βγει από την συμβαστική 27α και καλύπτεται στο 27β και αν ε, καταπέσει ψηφίζεται. Τα υπόλοιπα είναι σωστά, απλά θέλω να αφαιρεθεί από το 27α. Η τροπολογία 239 δεν θεωρώ πως καλύπτεται από τη συμβαστική πρόταση. Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη. Και δεύτερον, η τελευταία συμβαστική τροπολογία, υπαριθμών 54, είναι συμβαστική από δύο πολιτικές ομάδες, άρα ορισμού δεν είναι συμβαστική, είναι μια ενοποιημένη τροπολογία δύο πολιτικών ομάδων και αφορά μια τροπολογία της κυρίας Ποδηματά και μια τροπολογία του κυρίου Ρόντε, εμού και του κυρίου Χατζημαρκάκη. Αυτό είναι το, το κείμενο. Αυτό δεν συμφωνεί με την τροπολογία μας, δεν καλύπτει τα ίδια πράγματα, οπότε θέλω να φύγει από την ενοποιημένη τροπολογία και να ψηφιστεί χωριστά. Στο σημείο 54 που δεν θα πρέπει ούτως ή άλλως να λέγεται συμβιβαστική τροπολογία, γιατί προέρχεται από δύο ομάδες. Και εγώ δεν θέλω να είναι στην ενοποιημένη τροπολογία. Η 467 θέλω να ψηφιστεί χωριστά. Αυτό το έχουμε πει και στο παρελθόν και ελπίζω όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις να γίνεται σεβαστή η ε, επιθυμία της ομάδας μας. Ευχαριστώ. Gut, το σημειώνω, η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζαμε την ε, θέση της ε, κυρίας Εκ. Η γραμματεία το επαλήθευσε και είναι με συμβιβαστική τροπολογία εντός των κανόνων. Όσον αφορά τώρα το 27β, την τροπολογία, η τροπολογία της κυρίας ΕΚ είναι στο 27α και θα ψηφιστεί, άρα δεν υπάρχει ανάγκη να ψηφίσουμε χωριστά, να την ψηφίσουμε χωριστά. Ωραία. Ε, δεν, δεν θα κάνουμε συζήτηση τώρα. Να δούμε τι, τι θα ψηφίσουμε πρώτα απ' όλα. Ας ψηφίσουμε τι θα ψηφίσουμε. Υπάρχουν λοιπόν δύο προβλήματα. Θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση για το πώς θα προχωρήσουμε. Εάν θέλει να αποσύρει ή να ψηφιστεί μεμονωμένα κάποιος που έχει υποβάλει μια τροπολογία ή τροπολογία του, αλλά πρώτα απ' όλα μπορεί να γίνει αυτό, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αυτό δεν αποφασίζεται από την ε, πλειοψηφία και αποφασίζεται σύμφωνα με τους κανόνες. Συμβασικές τροπολογίες υπάρχει κανόνας από δύο ομάδες. Δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε για να το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, αλλά θα παραμείνετε, θα παραμείνετε λίγο παραπάνω. Έντσου, έχετε κάτι διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, δεν ε, μπόρεσα να βρω την ε, κάρτα μου για την ψηφοφορία, με συγχωρείτε. Έστειλα το... Μπορώ να στείλω τον το βοηθό μου να πάω να τη φέρει και εντωμεταξύ θα ψηφίζω δυνατά στους Ναι, ναι, κύριε Ρόντε, πρέπει να πω πως είναι απαράδεκτο σε μία... να σειρώμαστε σε μία συμβαστική τροπολογία χωρίς να έχουμε συμφωνήσει σε αυτήν. Δεν, γίνεται, δεν είναι δυνατόν δύο κόμματα να κάνουν συμβαστική τροπολογία και μετά όλοι οι υπόλοιποι να αναγκάζονται να την δεχτούν. Και αυτό έχει συμβεί εδώ πέρα στην 4.20, ε, στην 4.25 και στην 16. Α, όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν θέλω να να επαναλάβω γιατί είμαστε κατά, είναι, είναι σημαντικό για μας και ελπίζω λοιπόν τα... Να ακούστηκαν και τα, τα σχόλια της ε, κυρίας Εκ. Λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι. Και εμένα δεν με ρώτησε κανείς ε, και για τις συμβαστικές τροπολογίες, έτσι φαίνεται πως είναι ο κανόνας, αλλά Νομίζω εγώ όπως το αντιλαμβάνομαι μπορεί κάποιος να αποσύρει την δική του τροπολογία και ρώτησα την γραμματεία εγώ πρέπει να ακολουθήσω τους κανόνες. Οι κανόνες είναι πως δύο τροπολογίες από δύο ομάδες μπορούν να γίνουν μια συμβαστική τροπολογία. Το εάν είναι τώρα λογικό ή όχι ε, και εγώ δεν καταλαβαίνω όλους τους κανόνες δυστυχώς πρέπει να τους εφαρμόσω. Δεν ξέρω, ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα να ξεκαθαρίσουμε γενικότερα το τι γίνεται με τις ε, συμβαστικές αυτές ε, τροπολογίες. Γιατί και εγώ είχα κάποιες ε, εμπειρίες που ήταν κάπως περίεργες. Σήμερα, με πάση περιπτώσει, πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες όπως είναι και οπωσδήποτε θα λάβουμε υπόψη την παρατήρηση της κυρίας ΕΚ και την δική σας πως θέλετε να ψηφιστούν χωριστά οι δικές τροπολογίες. Οπωσδήποτε θα γίνει αυτό ξεκάθαρα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όχι, δεν μπορούμε. Τούρμες και η κυρία Ποδηματά. Οπότε, τεχνικά εδώ πέρα, στη συμβαστική τροπολογία 45 υπάρχουν δύο κόμματα. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες και οι φιλελεύθεροι. Οπότε, αν οι φιλελεύθεροι θέλουν να απομακρυνθούν από αυτή τη συμβαστική τροπολογία, έχει μείνει ένα κόμμα. Ένα κόμμα δεν είναι συμβαστική τροπολογία. Νομίζω πως η κυρία Εκ έχει δίκιο και ο κύριος Ρόντε. Αγαπητέ Κλοντ, κάθε κόμμα μπορεί να κάνει, να υποβάλει συμβαστικές τροπολογίες. Προϋπόθεση είναι δύο τροπολογίες από δύο διαφορετικά κόμματα. Α, αυτές υπάρχουν. δεν μπορώ να τα αλλάξω αυτό και δεν υπάρχει καμία διάταξη. Ε, Ζήτησα από την Γραμματεία να το ξεκαθαρίσει. Εάν υπάρχει κάποιος ε, κανόνας ε, που δεν θα επιτρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί το, το επιχείρημα είναι σαφές, με πείθει. Αλλά δεν είναι το θέμα το εάν με πείθει εμένα, αλλά ποιος είναι ο κανόνας. Θα εφαρμόσουμε τον κανόνα ως έχει. Και προφανώς εδώ πέρα κάτι πρέπει να βελτιωθεί στον κανονισμό. Κυρία Ποδηματά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ε, σε σχέση με τη συμβιβαστική τροπολογία 54, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Εκ, η συμβιβαστική τροπολογία 54 καλύπτει δύο συγκεκριμένες τροπολογίες. Την τροπολογία 426 που θα υποβάλει εγώ και την τροπολογία 427 της κυρίας Εκ, του κυρίου Ρόντα και του κυρίου Χατζημαρκάκη. Ένα θέμα είναι το τεχνικό, ποιοι είναι οι κανόνες, και ένα θέμα είναι το ουσιαστικό οι δύο αυτές τροπολογίες θεωρούμε και οι δύο πλευρές που έχουμε καταθέσει σχετικές τροπολογίες ότι δεν καλύπτεται η ουσία του στη συμβεβαστική 54 και γι' αυτό ζητούμε να τεθούν χωριστά σε ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνω μια παρατήρηση η οποία δεν είναι συνήθις. Αντιλαμβάνομαι τη διαφωνία πρώτον αλλά δεύτερον δεν είναι πρόβλημα γιατί ε, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά η πλειοψηφία δεν το θεωρεί ούτως ή άλλως ε, πρόβλημα. Τέλος πάντων, μπορούμε να συζητάμε τη διαδικασία μία εβδομάδα. Το καλύτερο νομίζω να ξεκινήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε με την συμβαστική τροπολογία 4. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Καλή αρχή. Προσέχετε να μην μου ξεφύγει τίποτα γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Περνάμε 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 και 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Όχι, συγγνώμη, κάτι ξέχασα. 45. Ευχαριστώ. 45 υπέρ. Κατά αποχές <clears throat> απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 σε 3 μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 σε δύο μέρη Δεύτερο μέρο υπέρ, κατά Αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά Αποχέ, εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά Αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά Αποχέ, εγκρίνεται. 150 και 151 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται να επαληθεύσουμε. 150 και 151 η ψηφοφορία. Εννέα παραπάνω από το ΕΛΚ. Δεν είναι δυνατόν. Θα ξεκινήσει ξανά η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ε, δεν, λειτουργεί το μηχάνημα. Μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος. Yeah, we count. We count. Ε, θα μετρήσουμε. Υπέρ των 150. Υπέρ παρακαλώ. Μήπως τώρα υπάρχει το ερώτημα αν ήταν παραπάνω από το ΕΛΚ. Μπορείτε, μπορούμε να του μετρήσουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι, εμένα λίγοι μου φαίνονται πάντως. Ε, εντάξει, ναι, με συγχωρείτε, αστείευτηκα. Τριάντα έναντι 19 και 6 εποχές. Δεν ξέρω. Ε, δεν σας κατάλαβα. Ναι, να, να, να κάνουμε την πρόσθεση. 34 συν 19 συν 6. Νο, κανονικά είμαστε λιγότεροι. Όχι, περισσότεροι. Can you tell it by micro? Perhaps you can tell it. Yes, uh, there are too many members. Eh υπάρχουν παραπάνω βουλευτές που ψηφίζουν από τα μέλη της Επιτροπής. Και, σύμφωνα με το μηχάνημα, όλοι τους είναι από το ΕΛΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η διαφορά 34 έναντι 19 είναι τόσο μεγάλη που δεν αλλάζει το γεγονός. Αλλά για τις επόμενες ψηφοφορίες 7, 7 μέλη του ΕΛΚ παραπάνω. Αλλά η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 7. Σύμφωνα με το μηχάνημα, ναι. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Συμφωνείτε να κάνουμε μια δοκιμαστική να δοκιμάσουμε το μηχάνημα. Λοιπόν, θα ξαναδοκιμάσουμε μία φορά με το μηχάνημα. Για, θα κάνουμε πάλι την ίδια ψηφοφορία. 150-151 ξεκινάει η ψηφοφορία. Έχουμε δύο ΕΛΚ και τέσσερις σοσιαλιστές παραπανήσιους. Παρακαλώ αφαιρέστε τους. Τέσσερις ΕΛΚ και δύο σοσιαλιστές μάλλον. Τρεις τώρα, δύο. Οι σοσιαλιστές είναι εντάξει και δύο ΕΛΚ περισσεύουν. Και πάλι ένας υπάρχει επιπλέον. Τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα ψηφίζουν 53. Μπορούμε λοιπόν να επαναλάβουμε την ψηφοφορία τώρα. Μόνο, τώρα θα ψηφίσουν μόνο αυτοί, όχι όλοι. Ξεκινάμε την ψηφοφορία για το 150 και 151. 53 ψήφισαν, 30 υπέρ, 21 κατά και δύο αποχές. Πολύ ωραία. Το αποτέλεσμα είναι σαφές, εγκρίθηκε με 31 ψήφους υπέρ. Παρακαλώ λοιπόν τώρα τις πολιτικές ομάδες να ψηφίζουν μόνο αυτοί που ψήφισαν και τώρα ώστε και τις επόμενες φορές να μην έχουμε προβλήματα. Ερχόμαστε στο 224. Ποιος ε, είναι υπέρ. Μάλλον ε, άρθρο 16α νέων η τροπολογία ΕΚ 224. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 154 καταπίπτει. Όχι όμως το 155. Ποιος είναι υπέρ. 155. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ μόνοι, ε, μόνο οι εξουσιοδοτημένοι για να ψηφίσουν. Εντάξει είμαστε. Λίγη ψηφοφορία. Ψήφισαν 51 και, και απερίφθη. 22 υπέρ, 25 κατά, 4 αποχές. Συμβιβαστική 18. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αν όλοι σηκώνετε σωστά το χέρι σας θα μπορείτε να μας το 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγη ψηφοφορία. Οι 24 υπέρ, 27 κατά απορρίπτεται. 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά Μπορώ να παρακαλέσω ποιος είναι υπέρ της 207. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Έλεγχος για τη 207 ξεκινά. Λίγη. Ένας ΕΛΚ ε, περισσεύει. Τώρα όμως είμαστε εντάξει. Λίγη ψηφοφορία. 30 υπέρ, 23 κατά, εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 συν 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Έλεγχος. Έλεγχος. Για την 24 συν 1 ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Απερίφθη. 212 υπέρ. Κοιτάζω με προσοχή λέει ο πρόεδρος ως επτοπλίστων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 32 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 27α υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 27α ξεκινά λίγη 28 υπέρ 23 κατά 2 αποχές εγκρίθηκε και καταπίπτει 27β και ερχόμαστε στην 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και έτσι ερχόμαστε στην 200 απε, ε, ε, συμβιβαστική 29 ψηφίζεται υπέρ κατά παρακαλώ και πάλι ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 262 και 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβεστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 264 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Συμβιβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 229 υπέρ κατά η 229 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 294 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 303 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβαστική 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 316 υπέρ κατά αποχές απορρίφθη 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τώρα έχουμε μία προφορική τροπολογία στην ε, τροπολογία 38 δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 42 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 200 242 ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά Λίγοι. Απερίφθη. 25 κατά, 24 υπέρ. Η τροπολογία συμβαστική 44 υπέρ. Με συγχωρείτε, κάτι μου, ε, μου ξέφυγε. Η 346 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 349 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές Παρακαλώ επαναλάβετε 349 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. <clears throat> Και τώρα έχουμε τη συμβαστική 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 363 υπέρ. Κατά δεν έχουμε ψηφίσει ακόμη και ζητάτε έλεγχο. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την ψηφοφορία. Νομίζω ότι καλό θα ήταν αν μπορούσαμε να δούμε τις, ε, την ψηφοφορία και των άλλων ομάδων και γι' αυτό ζητώ τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Κατευθείαν λοιπόν ε, την 363 ηλεκτρονικά. Λίγη. Λίγουμε. Ωραία. Είναι πολύ σαφές. 47 υπέρ, 5 κατά. Η 356 καταπίπτει. συμβιβασική 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 362 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 377 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος. Ο, ο θέλει πάντοτε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ξεκινά, λίγη. 22 υπέρ 30 κατά απερίφθη. Η 378 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. μετά καταπίπτουν όλες οι υπόλοιπες. Θέλει κανείς έλεγχο. Για την 378 δεν την κάναμε. Με συγχωρείτε, για την 378 ζητείτε ηλεκτρονικός έλεγχος, ξεκινάει. Ένας ΕΛΚ περισσεύει. Λίγοι. 38 υπέρ 10 κατά μία αποχή. Η ε, συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 389 νέα προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 390 υπέρ κατά και πάλι ε, ερωτήσεις σηκώστε το χέρι υπέρ για τις 390 κατά έλεγχος ηλεκτρονικός ξεκινά η ψηφοφορία 28 υπέρ 24 κατά εγκρίθηκε. 393 υπέρ. Επαναλαμβάνουμε τα αποτελέσματα της προηγουμένης ηλεκτρονικής 28 υπέρ 24 κατά. Ε, μπορείτε να ρωτάτε τη γραμματεία αν δεν με πιστεύετε. Ε, 393 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 404 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. 404 έλεγχος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίθηκε 26 υπέρ, 22 κατά δύο αποχές. Ε, η 404 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 405 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 407 κατέπεσε. Και ερχόμαστε στην βασική 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 412 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 413 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 417 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 420 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα με προφορική τροπολογία Ο κύριος Ρόντε. Ε, ε, δεν δέχομαι αυτή την προφορική τροπολογία διότι είναι μία προφορική τροπολογία στη δικιά μου τροπολογία και δεν συμφωνώ. Θα θέλαμε λοιπόν την αρχική μας τροπολογία 420 χωρίς την προφορική ε, επιπρόσθετη. Οπότε δεν επιτρέπεται αυτή η προφορική για να δούμε το μέλλον εάν μπορούμε να δεχθούμε στο μέλλον αυτή τη διαδικασία. Αν ένας διαφωνεί τότε ε, αποσύρεται η προφορική. Δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε υπό αυτά στις συνθήκες. Μπορείτε να καταγράψετε την ε, τροποποίηση τροπολογία στο κείμενο, από ό,τι μου είπε η Γραμματεία. Μπορεί να περάσει η τροπολογία δηλαδή στο καθεαυτό κείμενο. Um να είμαστε βέβαιοι. Βεβαίως ο κάθε εισηγητής μπορεί στην έκθεσή του να γράψει ε, τα συν και τα πλήν στον κατάλογο ψηφοφορίας. Αλλά μία προφορική τροπολογία όταν ένας διαφωνήσει ε, μπορεί να μην ε, βελτιώσει το κλίμα εδώ γιατί ο άλλος μπορεί να διαφωνήσει με το διαφωνούντα. Δυστυχώς δεν μπορώ να αλλάξω την διαδικασία άρα δεν μπορούμε πλέον Λοιπόν να ε, ψηφίσουμε την ε, τροπολογία αλλά ψηφίσουμε την αρχική 420 ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές <clears throat> κλείνει. εγκρίθηκε. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχέ ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 420 χωρίς την προφορική ε, τροπολογία. Απορρίπτεται. Κρίμας. Οι 425 σε δύο τμήματα και πάλι με το προφορική τροπολογίες. Με συγχωρείτε, πρώτα όμως έχουμε 422 του Γκίρεκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε 425 πρώτο και δεύτερο μέρος, απερίφθη η προφορική τροπολογία, άρα δεν ψηφίζεται και ψηφίζουμε την αρχικό πρώτο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές αποφασίζεται, υπέρ. Το δεύτερο μέρος, κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 54 που είναι το περίπλοκο θέμα και ψηφίζουμε. Και μετά τις μεμονωμένες. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής 54. Η κυρία Εκ. Όπως βλέπετε υπάρχουν δύο τροπολογίες, μία της κυρίας Προδηματά και μία δικιά μου, 426-427. Σαν ε, ολοκληρωμένη τροπολογία πρέπει να συμφωνήσω ότι αν ψηφίσουμε όπως λέει ο κατάλογος της ψηφοφορίας εγώ είμαι υπέρ του να ψηφίσουμε πρώτα την τροπολογία αποδηματά και μετά τις δικές μας διότι δεν θα θέλαμε της ε, τροπολογίας μας, ε, ε, την τροπολογία μας 427 να, είναι, να αποτελέσει μέρος της συμβιβαστικής 54. Δηλαδή αποσύρετε την δικιά σας τροπολογία, δεν σας κατάλαβα. Δηλαδή, τι θέλετε, θέλετε χωριστή τροπολογία, μου λέγονται ότι η συμβιβαστική είναι αποδεκτή, άρα ψηφίζουμε και δεν συζητούμε. Ή την αποσύρεται ή παραμένει. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα το οποίο με απασχολεί. Αν δύο άλλες ομάδες συμφωνήσουν και υπάρχει ε, μη ένα 50% για την ολοκληρωμένη τροπολογία δεν νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε την συμβιβαστική 54 διότι δεν νομίζουμε ότι το, το, το, κείμενο είναι το ίδιο και υπάρχει μία υφαρπαγή της δικιάς μου ή της δικιάς μας τροπολογίας. Το έχουμε ξανασυζητήσει στην αρχή της ημερησίας διατάξεως κυρία Εκ και εγώ μπορώ απλώς να σας πω τι βλέπω και τι καταλαβαίνω ότι η γραμματεία μου λέει ότι είναι δυνατόν να ψηφίσουμε τη συμβιβαστική, ίσως καλό θα ήταν να το διευκρινίσουμε γενικώ γιατί αντιλαμβάνουμε τις ε, ε, ε, τις ροπολογίες. Αποσύρετε την πρότασή σας κυρία Ποντιματά. Είστε από δύο μόνο τροπολογίες, τη δική μου και της κυρίας Έκ και του κυρίου Ρόντε. Εάν εμείς οι δύο που έχουμε υποβάλει αυτές τις δύο σχετικές τροπολογίες δεν καλυπτόμεθα από το συμβιβασμό. Εφόσον ο συμβιβασμός περιορίζεται σε αυτές τις δύο τροπολογίες, δεν υπάρχει συμβιβασμός κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να γίνει χωριστή ψηφοφορία. Το κατάλαβα το επιχείρημα. Μπορώ να σας πω από εκατοντάδες τροπολογίες που έχω καταθέσει πως ε, υπήρχε κάπου συμβαστική τροπολογία που εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν συμβαστική και κανέναν δεν είναι ενοχλούσε. Αυτή είναι η διαδικασία και εμένα μου φαίνεται περίεργη, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Και αυτή πρέπει να ακολουθήσω, λοιπόν. Αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό κατεπικόντως, γιατί εδώ πέρα δημιουργείται προηγούμενο που πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και τώρα θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία, δεν γίνεται αλλιώ και δεν θα το συζητήσουμε πλέον. 54 ψηφίζετε. Σας, σας παρακαλώ. Giles, ε, είναι, είναι απαραίτητο. Καλώς. Εσείς θα κρίνετε αν είναι απαραίτητο κύριε Πρόεδρε, αλλά πρέπει να πω... Ο συμβιβασμός των δύο ομάδων είναι μια τροπολογία, αποτελεί μια τροπολογία συμβιβασμού. Αυτό είναι γεγονός. Θα ήταν ατυχές εάν για τις άλλες τροπολογίες οι εισηγητές δεν είναι απόλυτα ευτυχείς, αλλά υπάρχει ο συμβασμός, Πρόεδρε. Ελπίζω αυτό να σας ικανοποιεί. Όξω όχι. ευτυχώς κάποιος με βοηθάει. Λοιπόν, κοιτάξτε, μπορούμε να, να, το συζητήσουμε, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες. Κύριε Χόλου, της διαδικασίας. Ελπίζω, να, μπορέσω να σας βοηθήσω κι εγώ. Δεν θα μπορούσατε να ακούσετε τις απόψεις των εισηγητών που λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το συμβασμό και θα το, θα το ψηφίσουμε ως προσθήκη. Το, ξεκι... το είπα στην αρχή πως πρώτα θα ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία και μετά τις δύο τροπολογίες, αν επιμένετε να ψηφιστούν. Αυτό, αυτό είπα να κάνω και νομίζω είναι με αρκετά καλή παραχώρηση. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 54. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της συμβαστικής 54. Κατά. Ε, θα επαληθεύσουμε αρχή ψηφοφορία. Πέρας. 26 υπέρ 25 κατά. Πάει αυτό. Και τώρα 426 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κοιτάξτε, ψηφίζουμε. Ναι, μπορείτε και να μην ψηφίσετε, είναι και αυτός ένας τρόπος. Αλλά έτσι πλέον δεν θα υπάρχει καμία πλούσια. Λοιπόν, 4.26 υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Αποχές. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ λέω πως το δεύτερο απορρίπτεται. 427. Να, να υπαλληθεύσουμε το δεύτερο της 426. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 4.27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. 427 άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 428 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Ε, καταπίπτει, συγγνώμη. 5 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ ξανά με συμβαστική τροπολογία σε δύο μέρη υπάρχει πάλι μια αντίρρηση στην προφορική τροπολογία, οπότε ψηφίζουμε το αρχικό χωρίς προφορική τροπολογία. 16, πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά απόχε. απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Α, να επαληθεύσουμε, αλλά ήταν ξεκάθαρο. Δεύτερο μέρος υπέρ. επαλήθευση. 16 δεύτερο μέρος, άρχη ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. Α, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο. Λοιπόν, συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 21ο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος αποσύρεται. 21 πρώτο μερος υπερ κατα κατά αποχές εγκρίνεται. Η 22 υπέρ 22 και 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται και περνάμε στην 6 της ίντα υπέρ Κύριε Τούρμες, δεν είδα την τροπολογία σας. Όχι. Την υπαριθμόν 2 και όχι ο συνάδελφος 2 βεβαίως. Η 2 του κυρίου Τούρμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τελειώσαμε. Όχι. 6 της ίντα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Α, καταπίπτει. 11 της ίντα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αυτό ήταν έχουμε και την συνολική ψηφοφορία. Δεν περίμενα να φτάσουν ως εδώ. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. <laughs> Είναι κάποιος παραπάνω από το ΕΛΚ. Και το αποτέλεσμα είναι 42 υπέρ, 3 κατά, τέσσερις εποχές, Συγχαρητήρια. Όλη καλή δουλειά. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία Τσίτσεστερ. Όχι, όχι άλλη συζήτηση, σας παρακαλώ. Κύριε Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Ναι, παρακαλώ για ένα λεπτάκι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις δεν είχα φτάσει σε τόσους συμβιβασμούς σε ολόκληρη τη ζωή μου. Έμαθα να φτάνω σε συμβιβασμούς, αλλά οι συμβιβασμοί έχουν πολλούς ορισμούς και αποχρώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Άντρου Χίλμαν, τη συνάδελφο και τη γραμματεία που με βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Oh, Λοιπόν, τώρα έχουμε την έκθεση Τσίτσεστερ. Κάποιες άλλες παρατηρήσεις ε, διαδικαστικές, κυρία Φανμπρέντ. Γνωρίζω ότι η, η έκθεση μου είναι πολύ ε, μικρή, γιατί έχει μόνο μία τροπολογία, αλλά νομίζω είναι πριν από την έκθεση Τσίτσεστερ. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ. Τόσο, τόσο χρόνο έχουμε αφιερώσει και παραλίγο να την προσπεράσουμε το αποτέλεσμα του ημερούς διαλόγου με την κυρία Φαν Την έχω συγχαρεί τρεις φορές, αλλά δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα. Λοιπόν, ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε. Τη κυρία Φαν Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Και πέρας και το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο. Συγχαρητήρια και πάλι και με συγχωρείτε. Τώρα περνάμε στην έκθεση Τσίτσεστερ. Συμβαστική 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σημείο. 2. Υπαριθμόν 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. να το ξαναπώ. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Α, όχι, 3 καταπίπτει. 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 σε 2 μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά απόχε εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 11 υπέρ κατά απόχέ απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 12 καταπίπτει 13 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ Α, συγγνώμη, ναι, δύο φορές το ίδιο είπα. Ε, πάνω από μία ώρα δεν τα καταφέρνω. 26 καταπίπτει, 27. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Και το αποτέλεσμα είναι εγκρίνεται σαφώς. Συγχαρητήρια. Περνάμε στην τελευταία ελπίζω ψηφοφορία καμία παρατήρηση, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε... Πρέπει να κάνουμε δύο ψηφοφορίε. Μία ψηφοφορία, κατευθείαν ηλεκτρονική, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Κάσπαρη και αυτό το τελευταίο κομμάτι σήμερα για τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ. Ε, δεν νομίζω συχνά να τις κάνουμε τόσο αναλυτικά τις ψηφοφορίες. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη, άμα βρω την ημερήσια διάταξη. Ja, ja. Also, noch Höchstwerte an Radioaktivität in Nahrungsmitteln und Futtermitteln im Falle eines nuklearen Unfalls und so weiter. Λοιπόν, ε, μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα δαριενέργεια και τα λοιπά. Εισηγητή ο κύριο Μπέλετ. Κυρίε και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Προσδεθείτε. Ησυχάστε για να μιλήσει ο κύριο Μπέλετ. Μόνο ο κύριο Μπέλετ. Ήβο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω Ολλανδικά, να κάνω την εισήγησή μου στα Ολλανδικά. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο αυτό έκθεση ακολουθεί μια πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατχήματος. Μιλάμε για αναδιατύπωση και πρέπει αμέσως να απογοητεύσω κάποιους που θεωρούν πως έχουμε μία σοβαρή αναδιατύπωση. Δεν συμβαίνει αυτό. Το περιεχόμενο των υφισταμένων κειμένων δεν αλλάζει. Όποιος έχει κάποια αμφιβολία να τον παραπέμψω στα έγγραφα που υπάρχουν στους ε, φακέλους μας. Στο σημείο 17 έχουμε μία επιστολή της ε, Νομικής ε, Επιτροπής και της Νομικής Υπηρεσίας και των τριών οργάνων Συμβουλίου, Κοινοβουλίου, Επιτροπής, οπότε δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία. Μιλάμε μόνο για μια κωδικοποίηση, κάτι το θεσμικό δηλαδή που αφορά τρεις κανονισμούς και οι οποίοι βεβαίω συγχωνεύονται. Ο λόγος λοιπόν είναι η προσθήκη ενός νέου εκτιμώντας, δηλαδή το εκτιμώντας 15. Και στην αιτιολογική αυτή σκέψη αναφέρουμε το γιατί έχει κάποιες αρμοδιότητες το Συμβούλιο. Δηλαδή αναφέρεται στο εκτιμώντας 15 πως λογικό είναι να διατηρεί το δικαίωμα εκτελεστικών εξουσιών για το Συμβούλιο. Οπότε έχουμε εδώ πέρα έναν μηχανισμό δύο βημάτων παρέμβασης σε περίπτωση στην οποία έχουμε κίνδυνο ακτινοβολίας από πενικό ατύχημα ή όπως αλλιώς προκύψει. Πρώτα απ' όλα υπάρχει καθήκον Κομισιόν να συντάξει έναν κανονισμό ad hoc για το συγκεκριμένο ατύχημα για τη συγκεκριμένη περιοχή και το συγκεκριμένο χρόνο, δηλαδή για συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, εάν ε, απελευθερωθεί η εκνοβολία. Το δεύτερο μέρος είναι πως εντός ενός μηνός από όταν ε, συνταχθεί αυτός ο οργανισμός ad hoc, το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τον κανονισμό της ε, Κομισιόν ή να τον μονιμοποιήσει. Οπότε δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία του κανονισμού, όπως σας είπα, αλλά έχω κάποιες ε, κριτικές ε, παρατηρήσεις παρόλα αυτά μετά από σύσκεψη με την νομική υπηρεσία. Εμείς θεωρούμε πως το εκτιμώντας το οποίο προστίθεται δεν ξεκαθαρίζεται γιατί υπάρχουν αυτές οι εκτελεστικές αρμοδιότητες οι οποίες δίνονται στο Συμβούλιο και επιπλέον θεωρούμε πως με το να χωρίζεται σε δύο φάσεις η διαδικασία όπου μπορεί να επιβεβαιώσει ή όχι τις απόφασεις Κομισιόν. Η δεύτερη αυτή φάση δεν έχει κάποια προσθέμενη αξία. Οπότε έχουμε κάποιες τροπολογίες που συνδέονται με το νέο αυτό εκτιμώντας 15, αλλά ε, βεβαίως έχουν κάποιες συνέπειες. Αυτό το οποίο προτείνω ως εισηγητής, όπως σας είπα σε συνεννόηση με την νομική υπηρεσία και αυτό το οποίο θα προτείνουμε ως Επιτροπή, είναι το εξής προτείνουμε να δοθούν στην Κομισιόν οι αρμοδιότητες σε περίπτωση ατυχήμενος να δράσει άμεσα για, τα, για την προσαρμογή των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων αδιενέργειας στο παράρτημα του κανονισμού και δεύτερον ζητάμε κάποιες ε, αρμοδιότητες, ζητάμε να οριστούν κάποιες αρμοδιότητες κάτω εξουσιοδότησης στην Κομισιόν για τα επίπεδα ε, ραδιενέργειας και τον κατάλογο τροφίμων για να μπορέσουν να αναθεωρηθούν όλα αυτά ε, και όλα αυτά να αποτελέσουν αρμοδιότητα της Κομισιόν. Η προσαρμογή δηλαδή των επιπέδων και ο το παράρτημα με τον κατάλογο των τροφίμων. για να λαμβάνει υπόψη νέες τεχνικές εξελίξεις. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση. Η δεύτερη πρόταση που επίσης προτείνουμε να αλλάξουμε και η τροπολογία εδώ πέρα είναι πως δεν θέλουμε μετά από πρόταση ενός αριθμού κρατών μελών να μπορούν να γίνουν αλλαγές. Δεν θεωρούμε πως κάτι τέτοιο είναι σωστό. Δεν είναι προς το συμφέρον της υγείας των καταναλωτών και θέλουμε να μείνουμε στις αρμοδιότητες της Κομισιόν και να μην πάνε σε έναν αριθμό κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή ο κανονισμός λέει μετά από πρόταση ενός αριθμού κρατών μελών. Αντί λοιπόν για αυτή την παρέμβαση σε δύο φάσεις, Κομισιόν και Συμβουλίου, ζητάμε στην περίπτωση ενός ποινικού ατυχήματος που μπορεί να είναι σε κάποιον αντιδραστήρα ή ξέρω εγώ μπορεί να είναι μια απελευθέρωση ακνοβολία σε ένα νοσοκομείο όπου υπάρχει πυρηνικό υλικό ή και σε άλλα μέρη προτείνουμε οι αρμοδιότητες της παρέμβασης να παραμείνουν στην Κομισιόν και ο κανονισμός και η ε, και θέλουμε οι εκτελεστικές αρμοδιότητες ε, του Συμβουλίου να καταργηθούν και να πάνε στην Κομισιόν. Και τέλος, όχι, πρώτο τελευταίο, Μιλάμε για το άρθρο 5 του κανονισμού. Μιλάμε για την πιθανή αναθεώρηση των ορίων της ακτινοβολίας, που είναι βεβαίως εξαιρετικά σημαντικό όπως αναφέρεται στο παράρτημα, η αρμοδιότητα για να αλλάξουν αυτά τα όρια σε περίπτωση νέας τεχνολογικής εξέλιξης ρητά να είναι στις αρμοδιότητες της Κομισιόν. Θα ήθελα να πω πως ε, το Συμβούλιο δεν θα έχει πλέον καμία αρμοδιότητα. Φαίνεται πως δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα, αλλά δεν ισχύει αυτό. Έχει την δυνατότητα να αποσύρει την αντιπροσωπεία αυτή και να την ενσωματώσει στο Συμβούλιο και βεβαίως μπορεί να μην ε, δεχτεί αυτές τις ε, αρμοδιότητες κατεξοδότηση. Μπορεί δηλαδή να τις ασκήσει το ίδιο. Οπότε έχει τον τελευταίο λόγο το Συμβούλιο. Τέλος, καταθέσαμε μία τροπολογία στο παράρτημα 1 που αφορά τον ορισμό της, των τροφών για μωρά που είναι σημαντικό και θέλουμε να το ευθυγραμμίσουμε με την νεότερη νομοθεσία γιατί εδώ πέρα αναφέρεται σε κείμενα της του 80. Οπότε ο νέος ορισμός αφορά δηλαδή το ποιες είναι μοριακές τροφές ε, είναι ε, παιδιά πρώτους ε, 4 με 6 μήνες της ζωής τους. Ενώ τώρα είναι τροφή για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 μηνών. Αυτός είναι ο ορισμός που βρίσκεται στο παράρτημα αυτού του κανονισμού. Οπότε μιλάμε για μια κωδικοποίηση, κύριε Πρόεδρε, ένα σημαντικό θεσμικό ζήτημα που θέλουμε να υπάρχει σαφήνεια για κάποιες εκτελεστικές αρμοδιότητες που θα εκχωρηθούν στην Κομισιόν, αλλά βεβαίως πάντα υπάρχει δυνατότητα αυτή η εκχώρηση να ανακληθεί από το Συμβούλιο, αλλά βεβαίως κατ' ουσίαν δεν αλλάζει τίποτα. Εάν έχουμε δηλαδή κάποιο ατύχημα ή απελευθέρωση ή ακτινοβολίας. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you. excuse me. Uh, Mr. Girek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni koledzy. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, γενικά συμφωνώ με τον εισηγητή. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο από πλευράς Επιτροπής πρόκειται για ένα αναμάσιμα παλαιών πληροφοριών. Γι' αυτό και δεν είμαι θετικά διακείμενος. Τα πυρηνικά τυχήματα, ιδιαίτερα το Τσερνομπίλ, μας οδηγούν στο να θέσουμε σωστές ε, προδιαγραφές ως προς τα ανώτατα επιτρεπτά όρια μόλυνσης ε, τροφίμων και Μετά το Τσερνομπίλ φτάσαμε σε μια κατάσταση ιστερίας. Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια μειώθηκαν δραστικά. Και δεν έλαβαν σωστά υπόψη τους ε, κανόνες που υπήρχαν τότε σε σχέση με την, τις θετικές μορφές ακτινοβολίας. Ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί είναι το εξής. 24 χρόνια μετά το ε, Τσερνομπίλ, το ε, κρέας ε, βοηδών δεν μπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρωπο διότι είχε ε, τραφεί παραδείγματο, ε, για, επί παραδείγματι με ένα είδος ε, μανιταριού. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι ο μέσος όρος ζωής ενός ισοτόπου ακτινοβολίας. Έχω πολύ σοβαρές ε, αμφιβολίες για τα παραρτήματα εδώ. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ε, υπάρχοντα επίπεδα. Και... Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα επίπεδα ε, ημιζωής που υπάρχουν και πώς εξελίσσονται. Δεν έχω καμία αμφιβολία σε σχέση με την νομική βάση, αλλά ε, έχω επιφυλάξει ως προς τα παραρτήματα 1, 2 και 3 που δεν λαμβάνουν υπόψη τα δικά μας ε, κριτήρια σε σχέση με τον υδροφόρο ορίζοντα, πώς μολύνεται μετά το Τσερνομπίλ και ούτω καθεξής. Αυτό αφορά τη στιγμή του ατυχήματος, αλλά και αρκετά αργότερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ακτινοβολία ως υπόβαθρο. Υπάρχει φυσική ακτινοβολία και θα πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέλετ για αυτή την εξαιρετική έκθεση και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ καταρχήν με τη δική του προσέγγιση για μία ενδοκινοτική προσέγγιση με την Επιτροπή Επικεφαλής ε, της Απόφασης των Επέδων Ακτινοβολίας παρά τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει ενιαία αγορά και οι ζωοτροφές εισάγονται και εξάγονται ελεύθερα στην Ευρώπη, νομίζω ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να προβάλλουν τα δικά τους ε, επίπεδα. Αυτό θα οδηγούσε στην ε, ολική καταστροφή. Νομίζω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιούν έτσι τα ατυχήματα για να προβάλλουν προστατευτικά μέτρα. Δεν μιλάω για μεγάλα ατυχήματα τα οποία είναι σαφή για όλους και όπου μιλάμε για υψηλά επίπεδα μόλυνσης, αλλά μπορεί να έχουμε να κάνουμε με ένα επιτόπιο ατύχημα και ορισμένα κράτη-μέλη θέλουν να αφήσουν ορισμένα προϊόντα εκτός αγοράς. Νομίζω λοιπόν ότι ενώ μιλάμε για ελεύθερη κυκλοφορία για ε, τις ζωοτροφές, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον εισηγητή και να αφήσουμε την Επιτροπή να αποφασίσει για τα επίπεδα. Επίσης ε, θα ήθελα να μιλήσω για την τροπολογία 2. Έχω μία υπόδειξη. Νομίζω ότι υπάρχει μία γραμμή που θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε. Γιατί ίσως έχουμε να κάνουμε με ένα πολυπολιτισμικό επίπεδο, πολύ περισσότερο από το 86. Γιατί νομίζω το, ότι το άμυλο θεωρείται ίσονο σημασία. Εδώ θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη και τα μπαχαρικά τα οποία χρησιμοποιούμε ε, λιγότερο, αλλά ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένα μπαχαρικά τα οποία χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο στην Αφρική ή σε ορισμένα μαγαζιά που ε, πολλούν αυτά τα μπαχαρικά, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες. Άρα θα πρέπει να δούμε τα προϊόντα ίσονος ή μίζωνος σημασία. Ε, κυρία Σαρτόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να φθηγραμμιστούμε κάπως, με τους συναδέλφους που έλαβαν τον λόγο πριν. Θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ευτυχή αυτό τον κανονισμό για να έχουμε μία κωδικοποίηση για το τι έχει επισυμβεί μέχρι τώρα. Δηλαδή να φτάσουμε σε μία κωδικοποίηση του status quo όμως είναι κάπως αποδυναμωμένη η πρόταση για το μέλλον. Δηλαδή δέχομαι το ότι θα πρέπει η Επιτροπή να φέρει το βάρος της απόφασης, λαμβάνοντας σε υπόψη ε, ένα ανώτερο επίπεδο παρέμβασης, ανάλογα με τον επίγοντα χαρακτήρα ατυχημάτων, λήψη αποφάσεων με βάση ατυχήματα. Αυτή η διαδικασία είναι θετική γιατί είναι μεταβατική. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό, δηλαδή κωδικοποιούμε, αλλά θα πρέπει να επινοήσουμε μια νέα στρατηγική. Διότι αυτά τα στοιχεία τα έχουμε κωδικοποιήσει με βάση τη μέχρι τούδε ε, πορεία μας, τόμας. Τούρμες, συγγνώμη, ο κύριος Τούρμες. Ε, καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την έκθεση. Ο Μισελ Ριβαζή θα δει τις λεπτομέρειες από τη δική μου ομάδα, γι' αυτό θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για την νομική βάση. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί καλύτερα στη δημόσια υγεία και την προστασία, την κοινωνική προστασία. Από ό,τι γιατί ζητάμε μία γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία για να δούμε πού θα εντάξουμε αυτή την ε, νομοθεσία. Όταν μιλάμε για κατεξουσιοδότηση πράξης, για εξουσιοδοτημένες πράξεις, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία εμείς ως Κοινοβούλιο χάνουμε αρμοδιότητες. Και στο τέλος μόνο το Συμβούλιο, μόνο το Συμβούλιο αποφασίζει, ελέγχει δηλαδή τη διαδικασία και κατά συνέπεια μπορούμε να έχουμε περίεργες αντιδράσεις, οι οποίες να μην είναι συντονισμένες μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς και, και του δίκαιου επιμερισμού. Άρα θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει μεγαλύτερο ρόλο και να είμαστε σίγουροι ότι δρούμε συντονισμένα. Ως προς το θέμα των υδάτων, Έχουμε μία ερώτηση προς την Επιτροπή. Διότι κατανοούμε ότι τα επίπεδα τριτίου και γενικής ακτινοβολίας καλύπτονται από ε, κάποιο άλλη, κάποια άλλη νομοθετική πράξη. Ως, ε, νομίζω ότι υπάρχει μία οδηγία για το πόσιμο νερό. Εάν η Επιτροπή λοιπόν μπορεί να μας εξηγήσει πώς αυτή η πρόταση της Επιτροπής μπορεί να ισχύσει και ευθυγραμμίζεται απόλυτα με αυτή την άλλη πράξη, τότε αυτό θα ήταν καλό. Γιατί δεν χρειάζεται ε, μία νομοθετική πράξη να έρχεται σε αντίφαση με μία άλλη τη στιγμή που τα κράτη-μέλη θέλουν να απομακρυνθούν από ορισμένες ε, οριακές τιμές οι οποίες ισχύουν για το πόσιμο νερό. Και ως προς τα επίπεδα υγείας και ακτινοβολίας ε, έχουμε αντιρρήσεις, αλλά νομίζω ότι ο συνάδελφος Ριβαζή θα τα δει σε λεπτομέρεια και θα σας αποστείλει τις παρατηρήσεις του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιζάρος. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή το 1987 πήρε μία απόφαση και σύμφωνα με αυτήν κάθε νομοθεσία πρέπει να κωδικοποιηθεί. Μέχρι στιγμής τρία θέματα που αναφέρονται στις οριακές τιμές ε, της ε, ακτινοβολίας στα τρόφιμα έχουν κωδικοποιηθεί και ουσιαστικά εδώ έχουμε μία περίληψη των τριών νομοθετημάτων και συμφωνώ με τον καθηγητή Γκέρεκ, δηλαδή συγχωνεύτηκαν τρία έγγραφα σε ένα και θα είχαμε ορισμένες επιφυλάξεις για το εάν πρέπει να εναρμονιστούν καλύτερα. Υπάρχουν πεπαλιωμένες παράγραφοι και επαναλαμβανόμενες παράγραφοι, οπότε αυτό δεν δίνει μια καλή εντύπωση όταν το εξετάζεται. Εξού και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον εισηγητή. Δεν βλέπω γιατί το Συμβούλιο θα έπρεπε ε, να έχει τέτοια ε, δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις. Πιστεύω ότι θα έπρεπε αντιθέτως η Επιτροπή να αποφασίζει και η εφαρμογή δηλαδή θα πρέπει να αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ τότε τους συναδέλφους. Ε, βλέπω ακόμη έναν ε, συνάδελφο που θέλει να λάβει τον λόγο. Θα μιλήσω Ολλανδικά κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα όμως πρώτα να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποθέτω ότι είναι εδώ κάποιος από την Επιτροπή, όχι τότε μπορούμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να έρθει την επόμενη φορά διότι ε, πολλοί ευρωβουλευτές έθεσαν ερωτήσεις στην Επιτροπή και εγώ θα ήθελα να θέσω ερωτήσεις και θα ήθελα προς το παρόν να κάνω ορισμένα σχόλια Ολλανδικά. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπε η κυρία Χολ και άλλοι συνάδελφοι για την κοινοτική μέθοδο. Νομίζω πως αυτή είναι η ουσία του πράγματος εδώ πέρα. Και πρώτα απ' όλα για τον κύριο Τούρμες οπωσδήποτε δεν θα κάνει κουμάντο το Συμβούλιο. Αντιθέτως, εάν δείτε τη τροπολογία, εμείς θέλουμε να κάνει κουμέντο η Κομισιόν, να μην διαλέξουμε δηλαδή τη διακυβερνητική, αλλά την κοινοτική μέθοδο, όπως ε, πολύ σωστά σύνοψε και η κυρία Χαλ, για να αποφύγουμε το ότι σε κάποια περιστατικά θα έχουμε καταστάσεις ε, προστατευτικές από κάποια Οπότε η Κομισιόν εδώ πέρα θα αποφασίζει γρήγορα και με τρόπο ευέλικτο οι προτάσει μεταξύ άλλων του καθηγητού Γκέρεκ και της ε, κυρίας Χολ και λοιπόν και του κυρίου Τούρμες για να παρέμβουμε στο παράρτημα του κανονισμού. Υπάρχουν τρία, τρία παράρτηματα. Το παράρτημα 1 μιλάει για τα επίπεδα για τα τρόφιμα, το παράρτημα 2 είναι ο κατάλογος των λεγόμενων ίσων σημασίας τροφίμων και έχουμε και το παράρτημα 3 που αφορά τα τις ζωοτροφές. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να κάνουμε κάποιες προτάσεις εκεί πέρα, να λέμε αυτό δεν είναι επίκαιρο, το τάδε πρέπει να αλλάξει. Αλλά το ερώτημα είναι με ποια νομική βάση θα γίνει αυτή. Εγώ θεωρώ πως δεν την έχουμε αυτή την νομική βάση. Το συνεννοήθηκα αυτό με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει νομική βάση, εκτός αν θέλουμε να δοκιμάσουμε για να στείλουμε ένα, ένα μήνυμα. Θα σας πω ότι μου είπε η νομική υπηρεσία, μου είπε πως με βάση τον ίδιο αυτό κανονισμό, ως κοινοβούλιο, το προσπαθήσαμε ήδη αυτό στο παρελθόν πριν από λίγα χρόνια και τότε έφτασε η υπόθεση στο δικαστήριο και εκεί πέρα χάσαμε την υπόθεση. Τώρα εντάξει μπορούμε να πούμε πως έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, νέα κατάσταση, αλλά επί της ουσίας δεν αλλάζει εδώ πέρα γιατί η Λισαβόνα δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ πέρα, μας το λέει η νομική υπηρεσία. Μπορούμε να κάνουμε μια νέα απόπειρα και να προσπαθήσουμε εκ νέου, όπως είπε ο κύριος Τούρμες, μέσω της δημόσιας υγείας και των νέων αρμοδιοτήτων που έχουμε εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει πως θα πάμε στην ε, συναπόφαση και θα πάει πάλι η υπόθεση στο 10, θα μας κοστίσει κάποιους μήνες και πιθανώς, ε, δηλαδή μιλάμε για 99 ή 95% πάλι όχι να μας πει, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε αν το επιθυμεί η Επιτροπή. Εγώ δεν είμαι υπέρ, βασίζομαι σε αυτά τα οποία μου είπε ως γνωμοδότηση η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Δεν λένε μην το κάνετε, αλλά είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να επιτύχουμε κάτι, γιατί υπάρχει ήδη ένα δεδικασμένο. Προσπαθήσαμε και επί δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ πέρα. Να πω και κάτι για αυτό το οποίο είπε η κυρία Σαρτόρη. Πώς κατ' ουσίαν μιλάμε για μια ενδιάμεση ε, κατάσταση και θα πρέπει στο μέλλον ε, να επανέλθουμε και να δούμε το πράγμα επί της ουσίας. Αυτά. Ε, νομίζω απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις και επίσης ε, και εγώ θα ήθελα να ζητήσω να είναι εδώ πέρα παρόντες οι της Κομισιόν επόμενη φορά. Μου λένε πως ο κύριος ε, Σιμαγκάλια είναι εδώ από την νομική υπηρεσία, μπορεί να απαντήσει. Συμφωνείτε? Εντάξει. είναι η σειρά σας. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη διότι καθυστέρησα. Ε, με συγχωρείτε. Θα ήθελα πολύ σύντομα να ε, σχολιάσω διάφορα θέματα που άπτονται ε, σε ερωτήματα που ετέθησαν για την αναδιατυπωμένη πρότασή μας σχετικά με τα ποσοστά ραδιοενεργής ε, ε, μόλυνσης των τροφίμων και των ζωοτροφών νομίζω ότι το μόνο σχόλιο το οποίο μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή επί του θέματος είναι ότι αφού διάβασα το σχέδιο της εκθέσεως που κατήρτισε η Επιτροπή αυτή θα ήθελα απλώς να τονίσω ότι με αυτήν την άσκηση κωδικοποίησης που η οποία έγινε ε, άσκηση αναδιατύπωσης ε, εξετάζουμε διάφορες διατάξεις εφαρμόσιμες αυτής ε, της, αυτών των κανονισμών αλλάζει το κείμενο του κανονισμού θα αντικατασταθεί και θα αρθεί για να υπάρξει ένας νέος κανονισμός. Στην αρχή θέλαμε να έχουμε ένα κωδικοποιημένο κείμενο, δηλαδή χωρίς αλλαγές όσον αφορά την ουσία. Αλλά ενώ διεξήγαμε την νομοθετική διαδικασία ε, σε σχέση με την αρχική κωδικοποιητική άσκησή μας διαπιστώσαμε μεταξύ τριών νομικών υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων ότι υπήρχαν επιφυλάξεις δυνατότητος εφαρμογής από το Συμβούλιο που δεν είχαν αιτιολογηθεί και σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μια τέτοια επιφύλαξη πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Εξού και χρειάστηκε να τροποποιήσουμε ε, την ε, άσκηση κωδικοποίησεως σε άσκηση αναδιατυπώσεως για να υπάρξει η προσθήκη του άρθρου 15 που ε, περιλαμβάνει την εισαγωγή της νέας διάταξης. Βέβαια στο σχεδιασμό έγιναν ορισμένες προτάσεις. Καλό θα ήταν η Επιτροπή Επιτροπής, ε, ε, οι υπηρεσίες Επιτροπής να αξιολογήσουν ε, αυτές τις προτάσεις για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε ουσιαστικές αλλαγές στην νομοθεσία αυτή. Αλλά φοβούμε πολύ ότι αυτή δεν είναι η μορφή με την οποία τέτοιες προτάσεις για αλλαγή μπορούν να συζητηθούν, διότι απλώς γίνεται μία κωδικοποίηση των ε, ισχυουσών ε, διατάξεων. Βέβαια, οι, οι υπεύθυνε υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να κληθούν, να εξετάσουν εάν μπορούν να ισχύσουν ορισμένες αλλαγές σε αυτή την νομοθεσία. Ατυχώς όμως όχι επί τη ευκαιρία αυτής της ε, αναδιατύπωσης της πρότασης. Είμαι διαθέσιμος για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση η οποία θα τεθεί σχετικά με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τούρμες έχει ζητήσει το λόγο. είχα θέσει συγκεκριμένες ερωτήσεις οι οποίες έπρεπε να τεθούν στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα όρια της οδηγίας ποσίμου ύδατος εάν δηλαδή υπάρχει ισότιμη μεταφορά και δεν έλαβα απάντηση καλό θα ήταν αν μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον εκπροσωπείται να μας δώσει μία απάντηση σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα. Από ό,τι γνωρίζω μπορώ, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα αλλά θα επανέλθουμε γραπτός με την απάντηση. Είσαστε ικανοποιημένος κύριε Τούρμες δεν είναι συνηθισμένο η Επιτροπή να παρίσταται και να μην μπορεί να απαντήσει αλλά αν δεν υπάρχει ο ειδικό, ελπίζω ότι την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε αυτό το θέμα ο αρμόδιος θα είναι στην αίθουσα. Ο κύριος Μπελέτ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον ε, κύριο Τούρμες όταν απαιτεί παρουσία της Επιτροπής. Ε, οπωσδήποτε. Αλλά αυτό το οποίο λένε εδώ πέρα οι νομικές υπηρεσίες νομίζω πως ε, εν μέρει αντικρούεται από αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ πέρα στο σημείο 17. Έχουμε επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων όπου αναφέρεται πως ε, εάν ε, η αρμόδια επιτροπή κρίνει πως ε, μπορούν, πως πρέπει να υποβάλει τροπολογίες θα πρέπει να ενημερώσει οπωσδήποτε Συμβούλιο και Κομισιόν. Αυτό το οποίο κάνουμε νομίζω εδώ πέρα με αυτό το σχέδιο έκθεσης εργαζόμαστε με βάση το άρθρο 31 της ε, συνθήκης Ευρατόμ, όπως έχει αυτή ενσωματωθεί η συνθήκη της ε, Λισαβόνας, δεν θέλω τέλος πάντων να τα κάνω αυτά δύσκολα, αλλά έχουμε κάποιες ε, συμβουλευτικές αρμοδιότητες, αλλά αυτό δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να υποβάλουμε τροπολογίες και αυτό βασίζεται σε μια επιστολή που έχουμε λάβει από τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου, που νομίζω αντικρούει αυτό το οποίο είπε ο αξιότιμος ειδικό ε, εδώ πέρα της νομικής υπηρεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι ε, η έκθεση σχετικά με την ανταγωνιστική πολιτική. Πρέπει να σας πω όμως προηγουμένως ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι ε, στις 8 Νοεμβρίου το μεσημέρι και τώρα ερχόμαστε στην έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 και δίνω το λόγο στην εισηγήτρια Σιλβάνα Κοχμερίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για δεύτερη φορά ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει αυτή την προσπάθεια δηλαδή η υπεύθυνη επιτροπή είναι η ΕΚΟΝ και εμείς γνωμοδοτούμε και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε από τις παραμέτρους έχουμε περιορισμένο χρόνο διότι ήδη μεθαύριο λίγη προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών όλα λοιπόν γίνονται πάρα πολύ γρήγορα Προσπάθησα ε, στην τροπολογία, ε, στην γνωμοδότηση αυτή να αναφερθώ εις ε, θέματα τα οποία απασχολούν και ουσιαστικά την Επιτροπή μας δηλαδή καταρχήν το θέμα της ενεργείας, το πακέτο απελευθέρωσης διότι υπάρχει ένα τρίτο πακέτο απελευθέρωσης και θα ήθελα να πιέσω ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το παρακολουθεί προσεκτικά και αντιστοίχως ε, να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και αν αυτό δεν βελτιώνει τις συνθήκες ανταγωνισμού να υπάρξει και πάλι ε, μία εκποίηση ε, του ενεργειακού τομέα. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα το οποίο εξετάζω είναι η συγκέντρωση μέσων ενημέρωσης. Ένα θέμα το οποίο ήδη είχε θίξει πέρυσι το κοινοβούλιο Κοινοβούλιο. Μέχρι στιγμής όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κοινοτοποιηθεί επαρκώς και θέλουμε να επανέλθουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τρόπο ώστε να μπορέσει να συμμορφωθεί στις προσδοκίες του Κοινοβουλίου. Τρίτον, η, τα τέλη για, την, για το roaming, ε, ε, δηλαδή ε, για την ε, ε, τις ε, τηλεφωνικές οι τηλεφωνικές διαλέξεις. Έχει μειωθεί η τιμή κατά 70% για τις ομιλίες και 60% για τα SMS. Παρόλα αυτά έχουμε ζητήσει να καταργηθεί τελείως ε, το τέλος ε, για την περιαγωγή, για το roaming και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα στο κείμενο. Δηλαδή ο ανταγωνισμός δεν επαρκεί στις αγορές αυτές. Αυτό διεπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σαν Επιτροπή ε, ε θέλουμε να διατυπώσουμε μια σχετική πρόταση. Μετά Μιλάμε για την ε, αύξηση των ε, συχνοτήτων ε, κινητής τηλεφωνίας όπου πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση αλλά είναι αδιαφανής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να μας πει πού έχει γίνει αυτή η πρόοδος, υπό ποιες προϋποθέσεις, ποιες χώρες θα εφαρμόσουν πόσο τις ρυθμίσεις και αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μία τόσο βασική πολιτική, για τόσο βασικά πολιτικό θέμα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν πλήρης διαφάνεια και ιδίω για μας τους βουλευτές να υπάρχει πλήρης πρόσβαση. Επίσης υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία τίθενται επανειλημμένως ε, και που έχουν απασχολήσει επανειλημμένως το Κοινοβούλιο, δηλαδή ε, να προσπαθήσουμε να δούμε αν τα θέματα αυτά ε, εφαρμόζουν τις διατάξεις διότι πολλά αλλάζουν και δεν είναι τόσο καλά οριοθετημένοι πλέον οι διάφοροι τομείς. Και τέλος το έκτο μου θέμα είναι ε, στη συνέχεια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητος να τονίσουμε και πάλι ότι τα διπλώματα ευραστεχνίας τα καινοτόμα είναι πολύ σημαντικά για τη βιομηχανία και πρέπει εντόνως να προσπαθήσουμε να υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα για διπλώματα ευρασιτεχνίας στην Ευρώπη και τέλος το σημείο το οποίο ήδη ε, αποτελεί ε, μία από πολλού χρόνου προειδοποίηση του Κοινοβουλίου προς ε, την Επιτροπή ότι δηλαδή θα πρέπει να συμπεριληφθούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να περιληφθούν στις διατάξεις αυτών των ρυθμίσεων. Αυτό είναι, έχω συζητήσει ήδη με ορισμένους ε, συντονιστές, με την κυρία Χέρτσοκ καταφέραμε να βρεθούμε βρεθούμε με άλλους είδα τους συνεργάτες τους αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συναντηθούμε κατά τρόπον ώστε να καλύψουμε όλα τα θέματα που μας απασχολούν σαν κοινοβούλιο και ε, να ε, κάνουμε μία γνωμοδότηση προς την ΕΚΟΝ που ασχολείται ιδίως με τις χρηματαγορές. Ευχαριστώ κυρία Κοχμερίν. Έχω δύο υποψήφιους ομιλητές στον κατάλογό μου. Πρώτα την κυρία Χέρτσοκ και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, συγχαρώ την εισηγήτρια για την εργασία της και γιατί έχει πρόθεση να συνεργαστεί με τους σκιώδεις ενεργά. Η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά το θέμα, δηλαδή να δούμε κατά πόσο οι κρατικές επιδοτήσεις βοηθούν πραγματικά τις ΜΜΕ. Συμφωνώ με όλα όσα είπε θα ε, ε, ε, έχουμε προετοιμάσει τις ε, τροπολογίες που έχουμε υποβάλει είναι συμπληρωματικές τροπολογίες. Καταρχήν χρειάζεται εξυγχρονισμός υποδομών ενέργειας και αυτό αφορά και τις επιδοτήσεις που θα πρέπει να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει να επισύρουμε την προσοχή της Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα άλλο ζήτημα που είναι μοναδικό είναι το εξής. Επειδή μιλάμε για κρατικές επιδοτήσεις λόγω κρίσης, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν ισχύει το ίδιο για τις καταστροφές, γιατί τότε δεν, γιατί δεν υπάρχει ειδικό ταμείο και ο μόνος ε, τρόπος βοήθειας της περιφέρειας είναι να δώσουμε μια κρατική επιδότηση ε, στην περίπτωση αυτών των επιχειρήσεων, όπως ισχύει με την κόκκινη λάσπη στην ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς οι κρατικές ε, επιδοτήσεις ε, είναι αναγκαίες σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλων καταστροφών. Αυτό ισχύει για την περίπτωση της Ουγγρα... Ουγγαρίας. Η τρίτη τροπολογία είναι να έχουμε οριζόντιες και εγκάρσιες πολιτικές. Η Telecom οι, οι τηλεπικοινωνίες μπαίνουν στο περιεχόμενο κάθε αυτό. Ε, πολλές φορές γίνεται συγχώνευση επιχειρήσεων και οι διαφορετικές πολιτικές επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων θα πρέπει να εξεταστούν εκ του, εκ του διότι οι συγχωνεύσεις επιταχύνονται. Αυτές είναι οι τροπολογίες και ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπένσον. Ευχαριστώ. Η γνωμοδότηση περιέχει σημαντικά ε, ε, θέματα ως προς την ουσία της εργασίας της Ήτρε. Θα πρέπει να γίνει σαφής ε, μνήα για το που βασίζουμε την πολιτική ανταγωνισμού, δηλαδή τις ανοιχτές αγορές και την ίση προσβασιμότητα και δίκαιη προσβασιμότητα για να υπάρχει αηφόρος ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Στο τομέα της ενέργειας νομίζω ότι αυτή η παράγραφος θα μπορούσε να ήταν πιο σαφής σε σχέση με τα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Επίσης, θα πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή να διασφαλίσει τον ανταγωνισμό στην ψηφιακή αγορά, όπου έχουμε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα, τις διαλειτουργικές προδιαγραφές ως προς τις ε. Πιστεύω ότι αυτή η παράγραφος θα πρέπει να ενισχυθεί. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε θα μιλήσει ίσως η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, η Κομισιόν καλωσορίζει το σχέδιο γνωμοδότησης, το οποίο κατά την απόψή μας για αρκετά σημαντικά ζητήματα. Βεβαίως, να υπενθυμίσουμε πως σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, με αυστηρό τρόπο είτε μιλάμε για κανόνες ανταγωνισμού, συγχωνεύσεων ή κρατικών ενισχύσεων. Προσέξαμε πως ακούστηκαν κάποιες εκκλήσεις για να χρησιμοποιήσουμε τα τομεακά μέσα έρευνας. Ε, τα σημειώνουμε αυτά, τα οποία είπε η συγγήτρια και ταυτόχρονα να υπενθυμίσουμε πως ε, θα χρησιμοποιηθεί το θα γίνει μια έρευνα για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα ατομιακά μέσα και θα πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το γενικότερο ζήτημα ή αν υπάρχει κάποιο ζήτημα ανταγωνισμού που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μέσα πολιτικής. Και εδώ πέρα αναφέρουμε στην αγορά της ενέργειας και τη συγκέντρωση των μημία των μέσων ενημέρωσης. Συμφωνούμε με την ανησυχία πως θα πρέπει να υπάρξει μια εσωτερική αγορά ενέργειας και σημειώνουμε τις ανησυχίες της συγγήτριας και τον γενικότερο στόχο που υπάρχει. Θα θέλαμε όμως να υπενθυμίσουμε αυτά τα οποία κάναμε πέρσι για να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Και πέρσι έχουμε λάβει και φέτος έχουμε λάβει κάποιες αποφάσεις ανταγωνισμού. Σε αυτή τη φάση σημειώνουμε τις ανησυχίες της ηγέτριας για την αγορά roaming και την, τον πληστηριασμό για τις συχνότητες ε, τέταρτης γενιάς κινητών και αυτό το οποίο είπε για το σύστημα έβρεση τεχνιών. Τέλος, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να υπενθυμίσουμε πως ήδη το 2009 προσπαθήσαμε να δώσουν περισσότερη έμφαση στις μικρόμεσες επιχειρήσεις ε, και στην έκθεση και νέα έκθεση την οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει να γράφουμε. Τέλος, κάτι άλλο συγκεκριμένα για τους σκιώδεις ηγητές όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Υπενθυμίζουμε πως δεν υπάρχει αλλαγή Συζητή τη Λισαβόνας για την συναπόφαση. Δεν ισχύει η συναπόφαση εδώ πέρα στον τομέα αυτόν, αλλά η Κομισιόν πάντα προσπαθεί να συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διάφορες προτάσεις και υπάρχει μια συνεχής ροή ε, εγγράφων όταν μιλάμε για διαβουλεύσεις σε διάφορες φάσεις. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια θέλει να επανέλθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Ναι, επειδή είναι σύντομος ο χρόνος, πιέζει. είναι σημαντικό να συνεργαστούμε έξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα αντικατοπτρίζει την άποψη της Επιτροπής. Θεωρώ πως και στις τροπολογίες που ανέφερε η Edith μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή γραμμή όσον αφορά την ενέργεια πακέτο απελευθέρωσης ενέργειας. Εδώ πέρα πρέπει να πούμε πως ακόμα και αν θεθεί εν ενέργεια το Μάρτιο του 2011 το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης πρέπει να δούμε εάν όντως βελτιώνονται οι συνθήκες του ανταγωνισμού και μετά πιθανώς να υπάρξει μια τομεακή έρευνα για μια γρήγορη εφαρμογή και αν δεν, εφαρμο... αν δεν βελτιωθούν γρήγορα οι συνθήκες τώρα, Οκτώβριο 2010, ε, αν το αναφερόμαστε στο 2009, είναι αρκετά έντονη η διατύπωση. Αν και επί της ουσίας συμφωνώ τώρα. Όσον αφορά τις αρχές, το κείμενο της πρότασης ε, νομίζω είναι πάρα πολύ σύντομο. Έχουμε 1500 λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, οπότε ε, έχω αναφέρει τις αρχές στις οποίες συμφωνούμε όλοι. Αλλά βεβαίως ε, μπορούν να κατατεθούν τροπολογίες για να προσθεθούν κάποιες αρχές. Δεν υπάρχει εκεί τόσος περιορισμός και νομίζω έτσι θα συμπληρώνονταν το κείμενο. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, μικρομεσαίες ε, επιχείρησεις και εκεί πέρα αν υπάρξει κάποια συγκλήρωση πάνω από τους 1500 ε, λέξεις νομίζω μπορεί να γίνει αυτό μέσω κάποιων τροπολογιών. Επίσης χαίρομαι και για τη συνεργασία που θα έχουμε με την Κομισιόν τα επόμενα χρόνια, γιατί ως Κοινοβούλιο μας ενδιαφέρει να έχουμε μια σωστή πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως υπογράμμισα και στην αρχή, μεθαύριο είναι η προθεσμία για τροπολογίες, οπότε αν θέλετε να καταθέσετε τροπολογίες πρέπει να βιαστείτε. Και μπορούν να κατευθούν τροπολογίες μόνο στα αγγλικά. Αυτά λοιπόν για το πρωινό κομμάτι της συνεδρίασής μας. Θα τα ξαναπούμε στις 3 η ώρα. Ευχαριστώ πολύ.